Dear colleagues, would you please take your seats? Okay, good afternoon everybody, dear colleagues. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Let's start our meeting. Να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση αυτής. Does it work now? Okay. To the point number one. Για ε, το σημείο 1 τη ημερήσια διάταξης, λοιπόν, έγκριση τη ημερήσια διάταξη θα ήθελα να κάνω τις εξή ανακοινώσει. Πρώτον, <clears throat> λόγω των διαπραγματεύσεων συμβιβαστικών τροπολογιών ε, και κάποιων άλλων τεχνικών ζητημάτων, η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών ζήτησε ε, να ε, αναβληθεί η ε, ψηφοφορία it's, it's, it's because of... μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ήταν μόνο για τεχνικούς λόγους, για να καταλάβω. Ε, όχι, λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπορούν να επιληθούν, λέει ο κύριος Βανίστελο, πριν από την ψηφοφορία. Είναι σχεδόν αδύνατο με ενημέρωσε μόλις η γραμματεία. Κρίμα, λέει ο κύριος Βανίστελ Μας ενημέρωσαν ότι ο κύριος Φελέγγι είναι άρρωστος. Ο κύριος Ιβάν Κόφκας θα τον αντικαταστήσει, που είναι ο, ε, ανα, ο ε, αναπληρωτής υπουργός ε, για, την, για τα εσωτερικά. Ο κύριος Βάγκαν, λοιπόν, είναι εδώ, Βόγκαν, και μπορούμε να αρχίσουμε με το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και αν συμφωνείτε όλοι θεωρούμε εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη και περνάμε στο 4. Όπως είπα, μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους σπόρους. Ο συντάκτης νομοδότησης είναι ο κύριος Ντέρεκ Βόγκαν και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για μια σύντομη παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω η παρουσίασή μου να είναι όσο το δυνατόν συντονότερη συντομότερη. Οι συνάδελφοι θα γνωρίζουν ότι είναι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας ε, για έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και είναι η πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων ε, για την γνωμοδότησή μας. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω το γεγονός ε, ότι η αποτελεσματική χρήση των πόρων είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία για την Ευρώπη 2020 και νομίζω ότι είναι σημαντικό τμήμα ε, της περιβαλλοντικής ε, ζωής ε, των Ευρωπαίων πολιτών και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητούμε αυτό το θέμα και που γνωμοδοτούμε από αυτού. Εξέφρασα εξ αρχής την σημασία των περιφερειών και των τοπικών αυτοδικήσεων ώστε να υπάρξουν σχέδια για την αποτελεσματική χρήση των πόρων νομίζω ότι οι περιφέρειες και τοπικές αρχές ε, πρέπει να ε, την χάνουν διαβούλευση κάθε φορά που λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις, γιατί κάθε περιφέρεια είναι διαφορετική και γι' αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη κατά την κατάρτιση των σχεδίων μας. Επίσης, αναφέρω στη γνωμοδότησή μου ότι εμείς ε, ως τοπικές αρχές δεν πρέπει να συμμετέχουμε μόνο στην κατάρτιση σχεδίων για τη βελτίωση ε, το, της χρήσης των πόρων ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικές αρχές και στην εφαρμογή, στην εκτέλεση αυτών των σχεδίων. Πολλές περιφέρειες και τοπικές αρχές ήδη συμμετέχουν στην εφαρμογή, στην εφαρμογή προγραμμάτων για την καλύτερη χρήση των ενεργειακών και υδάτινων πόρων ε, συμμετέχουν ε, όχι μόνο στην κατάρτιση, αλλά ήδη υπάρχουν και διάφορες συνέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στην Ουαλία, στη δική μου περιφέρεια, κάθε τοπική αρχή έχει ε, την, ε, το δικό της σχέδιο δράσης ε, για την χρήση των ενεργειακών πόρων και μάλιστα πρέπει να αποδεικνύει ότι προοδεύει ως προς την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Όσον αφορά τώρα τη χρήση των νέων τεχνολογιών και για τα απόβλητα και για τους ενεργειακούς πόρους πρέπει όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης να συμμετέχουν από το Ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι η βάση λοιπόν της σύντομης γνωμοδότησής μου. Ελπίζω οι συνάδελφοι να έχουν σχόλια και θα ήθελα να ενημερώσω και τους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 14η Ιουλίου. Μετά 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ε, και θα ε, ψηφιστεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος κάποια στιγμή τον Νοέμβριο. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η συζήτηση. Όσοι θέλουν να παρέμβουν, παρακαλώ. Ε, Από πλευρά σχεδόν εισηγητών, Ερμήνε Μαζόνη, δεν παρίσταται. Εσείς, παρακαλώ, εσείς. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ, ήθελα να συγχαρώ θα ήθελα να συγχαρώ για τη γνωμοδότηση αυτή των συντάκτη γνωμοδότησης και για την αποτελεσματική χρήση των πόρων που είναι το κλειδί για την αηφορία στην ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και αυτή η αηφορία στην ανάπτυξη θα πρέπει να είναι μία από τις κυριότερες ακριβώς κατευθύνσεις που θα αναλάβει η Πολωνική Προεδρία δεν περιορίζονται μόνο στα ορυκτά καύσιμα και το πετρέλαιο και άλλοι πόροι συμπεριλαμβάνουν τα τρόφιμα και το νερό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι οι περιφερειακές αρχές, οι περιφερειακές κυβερνήσεις που ο ρόλος τους τονίζεται από τον εισηγητή θα πρέπει να επικεντρωθούν στους τρόπους και μεθόδους για την χρήση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτών των πόρων πρέπει να σκεφτούμε και τι θα πρέπει να γίνει για την πιο αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων ώστε να περιοριστούν τα απόβλητα από πλευράς τροφίμων ή και ε, ε, υδάτων του νερού. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνει κατανοητό ότι κάποιοι από τους πόρους είναι πραγματικά πεπερασμένοι, είναι περιορισμένοι και πρέπει να τους διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Thank Σας ευχαριστώ, κυρία σρέντερ Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για το σχέδιο της γνωμοδότησης αυτό. Νομίζω βρίσκω ότι έχει αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία καλύπτει. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε κάποια σημεία που στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκουμε επίσης. Δηλαδή το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι είναι δυνατόν ήδη σε αυτήν την χρηματοοικονομική χρηματοδοτική περίοδο να υπάρξει προσαρμογή αλλαγή προγραμμάτων ώστε οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής να ληφθούν υπόψη. Αυτό το θεωρώ σημαντικό γιατί δίνει μια δυνατότητα αυτό και για τους Δήμους και κοινότητες και τις περιφέρειες να δοκιμάσουν κάποια πράγματα και να εξοικειωθούν με κάποια πράγματα λαμβάνοντας υπόψη την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο στήριξης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο πιστεύω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα θέματα τα συνδέει με οικονομικές ε, συνιστώσεις, με οικονομικές παραμέτρους. Η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας πρέπει να είναι σημαντικό σημείο για μας και αυτό δείχνει ποια σημασία έχει για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πράσινων θέσεων απασχόλησης. Το θέμα των τοπικών οικονομιών και περιφερειακών οικονομιών και των ευκαιριών για αυτές τις οικονομίες θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη διότι βλέπουμε ότι και στη Μεγάλη Βρετανία ε, μεγάλα προγράμματα ξεκινούν όπου και αποτελούν μέρος της εθνικής πολιτικής τους και αυτή την πτυχή πρέπει να την τονίσουμε και να τη συμπεριλάβουμε. Η τρίτη συνιστόσα, η τρίτη παράμετρος λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι δηλαδή το επίκεντρο επενδύσεων και δράσεων στην Ευρώπη θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι όλες οι πολιτικές θα στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην υπάρχει μια αντιτιθέμενη πολιτική, μια αντιφατική πολιτική όσον αφορά τις επενδύσεις π.χ. των διαθροτικών ταμείων. Και αυτή η πτυχή είναι σημαντική και πρέπει και αυτή να συμπεριληφθεί. Το βρίσκω καλό ότι ο εισηγητής τους διάφορους παίκτες ως εμπλεκόμενους τους αναφέρει και τους ονοματίζει Μπορούμε να το ενδυναμώσουμε αυτό. Μία ερώτηση έχω στο τέλος τέλος. Δεν είναι απόλυτος, απόλυτα σαφές στην τελευταία πρόταση στο σημείο 2. Τι σημαίνει αυτό όταν πολιτικές λέει αντιτίθενται η μία στην άλλη ε, ποια λύση προτείνει ο εισηγητής. Ε, αυτό θα ήθελα να το δούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σμιθ, παρακαλώ. Sanchez Schmidt. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω σύντομα στην σημασία της ε, περιφερειακής πολιτικής και της χρήσης των κονδυλίων. Είναι αποτελεσματική αυτή η χρήση κυρίως στον τομέα της ενέργειας και εγώ θυμίζω την τροποποίηση του κανονισμού ΦΕΝΤΕΡ για την αποτελεσματικό, ενεργειακή αποτελεσματικότητα της κοινωνικής κατοικίας. Επίσης ε, για την ε, διασυνοριακή και δαφική συνεργασία θέλω να πω ότι στα σύνορα εμείς μπορούμε αποτελεσματικότερα να στήσουμε στρατηγικές για τη διαχείριση των πόρων και πρόκειται για ένα μέρος όπου η συνεργασία είναι και πιο ζωντανή μεταξύ των γειτονικών χωρών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φαν Νίστερ Ρόι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον συντάκτη της νομοδότησης για το έργο του. Θέλω όμως να κάνω ένα βήμα πιο πίσω και να πω ότι ναι μεν στο παρελθόν στην Περιφερειακή Επιτροπή είχαμε συζητήσει για τη στρατηγική του 2020 για την Ευρώπη και πιστήσαμε με σαφήνεια ότι θέλουμε να υπάρχει μια υποχρέωση ώστε να καθορίζεται για τα κράτη-μέλη πώς τα αποκεντρωμένα επίπεδα θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Και τότε όσον αφορά μια συμμαχία ή ένα συνασπισμό περιφερειών είχαμε κάνει λόγο. Τώρα η Ευρώπη θα πρέπει να παρέμβει σε αυτό, διότι στα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθοριστεί πώς οι περιφέρειες και τα αστικά κέντρα θα συμμετέχουν. Δεν γίνεται φυσικά όλα να τα καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι και να είναι όλα μεταβλητά. Υπάρχουν κάποιες ναυαρχίδες, κάποια, κάποιες ιδιαίτερες πρωτοβουλίες και σε σχέση με αυτές ε, για τη συμμετοχή των περιφερειών για αυτές τις ναυαρχίδες πρέπει αυτές οι γενικές παρατηρήσεις να ισχύουν ότι για παράδειγμα θα πρέπει να συμμετέχουν οι περιφέρειες. Και το Συμβούλιο τέθηκε θετικά όσον αφορά τους μηχανισμούς για τις πρωτοβουλίες αυτών των ναυαρχίδων της στρατηγικής μας. Και ο ρόλος των περιφερειών πρέπει να τονίζεται. Θα πρέπει να λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι μια προϋπόθεση ως αναγκαία συνθήκη να καθορίζεται από τα κράτη-μέλη πώς οι δραστηριότητες αυτών των ναυαρχίδων θα υλοποιούνται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ματσόνη είναι η συγγήτρια, σκιώδης η συγγήτρια του ΕΛΚ. Θα προσέλθει με κάποια καθυστέρηση πιο ύστερα. είπε όμως ότι μπορεί να προσυπογράψει αυτούς τους στόχους. Θα ήθελα να πω δύο λόγια και για το Περιφερειακό Ταμείο και τα κονδύλια του. Στις περιφέρειες πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις και στα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις. Τώρα, για το ότι αυτό θα είναι, λέει, στόχος, πρέπει στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές. Τίθεται το ερώτημα, πώς τα αστικά κέντρα και οι περιφέρειες θα μπορούν να διασυνδέονται με αυτούς τους στόχους. Τα αστικά κέντρα και οι περιφέρειες θέλουν να συμμετέχουν όχι μόνο στην εκτέλεση, αλλά και στο σχεδιασμό. Σχεδιασμός λοιπόν και εκτέλεση βαίνουν εκ παραλίλου και γι' αυτό αυτά τα βήματα πρέπει να γίνονται από κοινού και να βαίνουν παράλληλα. Ένα άλλο σημείο τώρα για κάτι το οποίο λειτουργήσε καλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη για τον κανονισμό για την αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας έχει κάνει λόγο για τις πόλεις. 164 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεν είναι αυτά επιδοτήσεις ή ε, χορηγίες αλλά δάνεια. Και υπάρχει μεγάλο περιθώριο εδώ, διότι με τράπεζες, με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γίνεται λόγος για την χρήση καινοτόμων ε, χρηματοοικονομικών μέσων. Πιστεύω καλά θετικά εργαλεία πρέπει να έχουν οι πόλεις ε, και οι περιφέρειες στη διάθεσή τους. Σημαντικό είναι να δημιουργηθούν όμως οι προϋποθέσεις γι' αυτό και θα καταθέσω και τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Βλάσεκ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ορισμένα πράγματα τα οποία είπαν ήδη και άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητος ο συντονισμός ε, σε διάφορα μεμονωμένα επίπεδα. Στο τοπικό επίπεδο, στο περιφερειακό, και βεβαίως και σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά τα επίπεδα πρέπει να διασυνδέονται. Υπάρχει επίσης και η διασυνοριακή συνεργασία και αυτή πρέπει να βελτιωθεί. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε τη δικτύωση. Αν παράγουμε ενέργεια, και πρέπει να, τη μεταφέρουμε, πρέπει να κάπως στον τόπο χρήσης της και δεν πρέπει να μας διαφεύγει και αυτό το σημείο. Okay, thank you very... Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Βόγκαν στη σημασία που δίνει για την ε, ε, για το πόσο σημαντικές είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, για το θέμα αυτό. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διεξάγεται πολιτική και σε τοπικό επίπεδο και αν θέλουμε πράγματι να είμαστε αποτελεσματικό, αποτελεσματικοί σε τοπικό επίπεδο, στους τοπικούς φορείς, πρέπει όλοι οι φορείς να συμμετέχουν προς ένα κοινό συμφέρον. Το, τα προβλήματα βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλα γιατί η Ευρώπη του 2020 και η σχετική στρατηγική θα μας πάει πολύ πέρα από το 2020 μέχρι το 2030, 40 μέχρι τότε θα έχουμε όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό, θα έχουμε πολύ περισσότερες ανάγκες ενεργειακές και οι τρέχουσες τάσεις, σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις ε, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και σε αύξηση πληθυσμού 19 δισεκατομμυρίων. Οπότε λοιπόν, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα ήδη με τον πληθυσμό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν ε, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν στη διαδικασία γιατί θα πρέπει να υπάρξει κάποια πολιτική πολύ συγκεκριμένη, ενδεχομένως ε, νέες τεχνολογίες ε, να ε, σχεδιάζονται σε κεντρικό επίπεδο, όμως πρέπει να γίνεται η διάδοσή τους και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να συμμετέχουν οι τοπικές αρχές, ώστε να, μπορούμε, να μπορούν να συμμετέχουν και στις πολιτικές ε, στόχο, αλλά και στην εφαρμογή. Και στην εφαρμογή πρέπει να συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό, γιατί έτσι θα έχουμε μια πιο συντονισμένη ε, προσέγγιση και θα έχουμε μια καλύτερη αίσθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του που πηγαίνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε, προ... είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίβερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ο συντάκτη νομοδοτήσης σωστά τονίζει στην πρότασή του ότι τα περιφερειακά κονδύλια σε αυτόν τον ρόλο διαδραματίζουν ένα κέριο ρόλο, ιδιαίτερα σημαντικό. Και αυτό ο ρόλο μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων τη στρατηγική 2020 διότι η αποδοτικότητα των πόρων διαδραματίζει ένα κέριο, κεντρικό ρόλο. Πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε κατά πόσον θα δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα επικυρώνονται μεγαλύτερα τέτοια σχέδια και προγράμματα, τα περιφερειακά και άλλα προγράμματα, να προσέχει ιδιαίτερα την συνιστόσα, την παράμετρο της αποδοτικότητας των πόρων ώστε <clears throat> να ζητείται από τα κράτη-μέλη επιπρόσθετα να δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Οι περιφέρειες και οι δήμοι και οι κοινότητες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο ήδη στο σημερινό υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όσον αφορά την ε, υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Ας σκεφτούμε τα απόβλητα, όπου οι δήμοι και κοινότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αποκομιδή ε, των αποβλήτων, των σκουπιδιών. Εδώ μπορούμε να προσπαθήσουμε τις λύσεις σε σχέση με τα επιμέρους κράτη-μέλη που βρέθηκαν για δήμους κοινότητες ε, να τονίσουμε αυτές τις πτυχές. Γι' αυτό αξίζει ο προβληματισμός, να δούμε οι βέλτιστες πρακτικές ως δίκτυο, ως network ε, των best practices δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω δήμων κοινοτήτων ώστε οι καλύτερες λύσεις να ε, μιμηθούν, να μιμηθούν άλλοι και να αντιγράψουν τις καλύτερες λύσεις όχι μόνο στα απόβλητα αλλά και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και έτσι να μπορέσουν οι περιφέρειες να συνεργαστούν με άλλους που έχουν δυσκολίες για την επίτευξη των στόχων. Έτσι θα μπορούσαμε με αυτή την αμοιβαία διαδικασία εκμάθησης να πετύχουμε πολλά πράγματα και θα καταλήγαμε προς την κατεύθυνση της αποδοτικότητας των πόρων. Θα ανακουφίζαμε την Ευρώπη Πιστεύω ότι πολλές λύσεις σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο μπορούν να εξευρεθούν με υποδειγματικό χαρακτήρα. Οι γνώσεις όμως έχουν πολύ μικρή διάδοση και δεν έχουν διαδοθεί επαρκώς και γι' αυτό θα πρέπει αυτή η παράμετρος να προαχθεί. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Σμόλκοβα. Ευχαριστώ πολύ. na to, čo je dôležité pre efektívne využívanie zdrojov. To je regionálna a miestna úroveň. Μικροφωνίζει έντονα και δεν μπορούμε να ακούσουμε τη διερμηνία από την ομιλήτρια. Μικροφωνισμός τρομερός. Zatiaľ čerpe z fondových prostriedkov. Excuse me for interrupting you. the interpreters have enormous problems, please. Počujete ma? Áno, môžem. No. Μικροφωνίζει διαρκώς και δεν μπορούμε να ακούσουμε παρότι ομιλεί από το μικρόφωνο. Α, οκ. Βημένη μικρόφωνο. Počujete ma? Môžem? Počujete ma? Môžem? Nie? Mám mikrofón. Έχω τώρα το μικρόφωνο, με ακούτε? Nie. Haló? Sorry. Nie, nie, halo. Nie počuť. Translate. Počuť? Môžem? Yeah, you can μπορούμε να ακούσουμε καλά την ε, Ευρωβουλευτή. Δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα όταν ομιλεί. Το πρόβλημα υπήρχε από τη διερμηνία αυτών που έλεγε, από την άλλη καμπίνα. Εντάξει, Τώρα είναι εντάξει για τα σημεία 4 και 5. Αυτό που είναι σημαντικό για την ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων και βλέπουμε ότι αυτό εμπλέκει το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δήμους και κοινότητες και έχουμε και στατιστικά στοιχεία από τη δική μου χώρα, από τη Σλοβακία που καταδεικνύουν ότι η Σλοβακία δαπανούσε μόνο 18,5% από αυτό το, ε, την περίοδο και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να είμαστε από τους πρώτους και όχι από τους τελευταίους. Πρέπει να καταφέρουμε να αυξήσουμε αυτή την συμμετοχή. Το τοπικό επίπεδο και το περιφερειακό επίπεδο δεν συμμετέχει επαρκώς. Στο σημείο 5 λοιπόν της ε, γνωμοδότησης που συνιστά τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν συστάσεις και προτάσεις και μέτρα για την συμμετοχή των εθνικών επιπέδων διοίκησης ε, και των περιφερειών είναι πολύ σημαντική υπόθεση και πρέπει να υποστηριχθεί. Okay, thank you very much. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κύριε Μοσέρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζουμε όλος ιδιαίτερος ε, την ανταπόκριση της Επιτροπής σας. Θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερος ε, την ε, σημασία της έντονης συμμετοχής όλων των επιπέδων της διακυβέρνησης και της τοπικής και της περιφερειακής. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι οι τομείς πολιτικής είναι πάρα πολύ και επιτάσσουν την συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ε, πολιτών και βεβαίως και των ε, πόλεων, ε, των δήμων και των κοινοτήτων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αποτελεσματικά λαμβάνονται οι αποφάσεις, ότι υπάρχει εφαρμογή των χώρων σχεδίων ε, τα, ε, το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο μόνο το ευρύτερο πλαίσιο μπορούν ε, να προσφέρουν, να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα, όπως για παράδειγμα σωστές τιμές, εξασφάλιση του, γεγονότη, του γεγονότος ότι απαγορεύονται κάποιες επιβλαβείς ουσίες ή περιορίζεται η χρήση τους, αλλά το πώς θα γίνει αυτό και το ότι θα γίνει κάτι τέτοιο βέβαια είναι ε, κάτι που εξετάζεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο ε, είναι το Συμβούλιο των Δημάρχων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια διαδικασία που έχει διερευνηθεί. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να, διερευνηθεί, να διευρυνθεί αυτή η ε, διαδικασία για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν ας πούμε ε, με τους ενεργειακούς πόρους όπως η βιοπικιλότητα πέρα από το θέμα της ενέργειας, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, της εποχής μας. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια και βέβαια οι δήμαρχοι έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, μπορούν να ενισχυθεί όμως περισσότερο ο ρόλος τους και μπορεί να χρειαστεί κιόλας κατά τα ερχόμενα έτη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ε, πρότεινε μία ενεργειακή οδηγία μια οδηγία για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας την οποία θα διαπραγματευτούμε στην αρχή ε, του ε, επόμενου έτους, τέλος του τρέχοντος και αρχή του επόμενου έτους και βεβαίως ε, ευχαρίστως θα δεχθούμε και τη δική σας υποστήριξη γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο να περάσει ο καιρός. Η ενέργεια είναι ένας από τους αμεσόδερους τρόπους να εξασφαλίζει κανείς για να έχουμε μάλλον όσο το δυνατόν καλύτερη ενεργειακή αυτονομία πρέπει να μειώσουμε όσο το δυνατόν τις εισαγωγές μας, πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αυτάρκεις. Ε, ε, βεβαίως έχουμε προβεί σε διαβουλεύσεις, ε, έχετε και εσείς πολλές φορές γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό, μιλώντας όλος ιδιαίτερος για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και έχετε εκφραστεί πολύ θετικά σε σχέση με, το, με τις πρωτοβουλίες που έχουμε προτείνει. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες έξι εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Οι υπόλοιπες αφορούν ένα-δύο τομείς πολιτικής, όμως η συγκεκριμένη αφορά δέκα διαφορετικούς τομείς πολιτικής, τη γεωργία, την αλληλεία, τις κλιματικές περιβαλλοντικές αλλαγές, μεταφορές, ενεργειακή πολιτική και βεβαίως και την περιφερειακή πολιτική. Ένα ζήτημα που αφορά όλους τους τομείς της ε, πολιτικής. Η περιφερειακή πολιτική θα είναι, από τις, μια ε, από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης. γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει και... Ε, να μην υπάρχουν αντιβάσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μέσων. Είναι καλό λοιπόν να υπάρχει μια ε, καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, με τα κρατημέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν όλα όπως πρέπει και βέβαια να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ιδεών ώστε να εντοπιστούν οι καλύτερες ιδέες για να επιτύχουμε του στόχους μας. Επίσης προτείναμε μια αναθεώρηση του προπολογισμού στις 29 Ιουνίου. Πρέπει να έχουμε και μια συγκεκριμένη πρόταση ειδικά για την περιφερειακή πολιτική και θέλουμε να δώσουμε τα απαραίτητα κριτήρια ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση που έχουμε, που είναι δύσκολο να την ε, βρούμε ειδικότερα σε περίοδο κρίσεω, ε, να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι η χρηματοδότηση αυτή θα δαπανάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι εκπληρώνει συγκεκριμένου στόχου ε, και σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ενεργειακής αποτελεσματικότητας και για ζητήματα μεταφορών και βιοπικιλότητας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι στόχοι θα εκπληρωθούν. Περιμένουμε λοιπόν ε, εναγωνίως να συνεργαστούμε μαζί σας ε, αλλά και με συναδέλφους σας σε, άλλους πολιτικούς σε άλλες επιτροπές γιατί πολλές είναι οι επιτροπές ε, τις οποίες αφορά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει και αυτό τον αντίκτυπο. Πρέπει να δούμε πώς θα προετοιμάσουμε τις πολιτικές αυτές, πώς θα τις σχεδιάσουμε, αλλά πρέπει επίσης να τις αξιολογήσουμε τις πολιτικές μετά. Όλοι οι φορείς πρέπει να συμμετέχουν, ε, πρέπει να απευθυνθούμε και στους πολίτες, να τους εξηγήσουμε γιατί θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και επίσης να τους εξηγήσουμε και ποιο είναι το κέρδος από όλη αυτή τη ε, ε, διαδικασία. Βέβαια, εντάξει, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που, για τα οποία πρέπει να επαναχωρήσουμε. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Δεν είναι δυνατόν να τα ε, καταφέρουμε όλα. Μερικές φορές πρέπει ε, να αφήσουμε πίσω κάποιους στόχους για να ευνοήσουμε κάποιους άλλους. Ελπίζουμε όμως ότι θα συμφωνήσει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τη για τη συζήτηση. Ο κύριος Τέρεκ Βόγκαν τώρα, ο εισηγητής, ε, θέλει να πάρει το λόγο για να κάνει τις τελικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για τις ε, προτάσεις τους και συνεισφορές τους. Σε όλες αυτές ε, με πολύ λίγα διαφωνώ και σχεδόν πρέπει να πω βρίσκω ότι όλα όσα είπα να έχουν νόημα και μπορούν να γίνουν δεκτά. Ο πρώτος ομιλητής έθιξε κάποια σημαντικά θέματα δεν κάνουμε μόνο λόγο για τα θέματα το, τα ενεργειακά και το νερό, αλλά και τα τρόφιμα, τα ορυκτά και πολλά άλλα ως παραδείγματα σημαντικές παρατηρήσεις ε, και ίσως επειδή δεν το ανέφερα, ίσως στις εισαγωγικέ παρατηρήσεις μου, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και διαχείρισης πρέπει να εμπλέκονται πάντα οι πολίτες ε, σε όλα τα επίπεδα ώστε αυτό να μπορεί να τονίζεται από πλευράς και της γνωμοδότησης όπως πρέπει δεόντως και για τη δεύτερη, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη παύλα, εκεί όπου αναφέρονται τα ωφέλη που πρέπει να υπάρχουν, trade-offs και νομίζω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπήρξε τοποθέτηση και για τις διαφορετικές τριβές ή ε, σημεία τριβών που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση για κονδύλια, για προγράμματα μεταφορών. Πολλές φορές ε, μπορεί να αισθάνονται κάποιοι ότι υπάρχουν ε, αντιτιθέμενοι, αντιπαρατιθέμενοι στόχοι και εδώ θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σε βάθος ε, για να δούμε τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη να μπορέσουν έτσι να προσαρμοστούν τα υφιστάμενα προγράμματα ώστε να επιτευχθεί η αποδοτικότητα των πόρων. Πρέπει να εντάξουμε στις ε, πολιτικές μας ε, και τις πολιτικές για την προστασία του κλίματος στο mainstreaming αυτό. Είναι σημαντικό για το μέλλον, στη στρατηγική 2020, αλλά επίσης και για την τα πολυετή χρηματοοικονομικά πλαίσια ε, multi-annual financial programs αυτά πρέπει να δούμε και πόσα από τα διαθωτικά κονδύλια θα μπορέσουμε να πετύχουμε βέλτιστη αποδοτικότητα. Ένα παράδειγμα που είδα όταν ε, προσπάθησα να δω σε σχέση με την Πολωνία και με τον συνάδελφο Βότσεκ για, την, ε, ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την, ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια βρίσκονται σε καλή πορεία. Πρέπει αυτά τα παραδείγματα να πάρουμε και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε ως βέλτιστες πρακτικές από αυτά να μάθουμε από αυτά που γίνονται στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ε, σημαντική παρατήρηση του κυρίου Φανίστελ Ρόι για την ανάγκη να εμπλέκονται οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές όχι μόνο στο υποόρους βέλτισης ε, διαχείρισης αλλά και σε σχέση με τις προσαρμογές. Το αναφέραμε αυτό όσον αφορά την έκθεσή μας ε, και όταν τονίσαμε ότι προτείνει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει ένα δίκτυο θα πρέπει όμως να εμείνουμε και να επιμείνουμε οι τοπικές αρχές και οι περιφέρειες να εμπλέκονται πλήρως ε, στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση. Έχουμε υποσχέσεις ε, που δίνονται αλλά πρέπει να υλοποιούνται. Πρέπει να βρούμε ένα πιο επίσημο τρόπο, ένα μηχανισμό επισημοποιημένο που θα μπορέσει να λειτουργήσει ώστε όχι μόνο για την πολιτική συνοχή αλλά και για άλλες ε, πολιτικές για τη βέλτιστη χρήση με αποδοτικότητα των πόρων. Με αυτές τις παρατηρήσεις θέλω να πω ότι έκαναν ενδιαφέρον ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και σχόλια οι συνάδελφοι και με αυτές τις ε, τροπολογίες που θα κατατεθούν αυτές θα πρέπει να είναι οι προτάσεις. Ευχαριστώ. 14 Ιουλίου, 12 η ώρα το μεσημέρι, είναι η προθεσμία για την ε, κατάθεση τροπολογιών. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμό 5, η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012, όπω τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, όλα τα τμήματα. Κύριε Σουριαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μιλήσω για τρία πράγματα. Καταρχήν, να δούμε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης τι έχουμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού από την Κομισιόν και να, να πούμε τι, σε τι δίνουμε εμείς τις ευλογίες μας. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε θέση σε αυτό που προτείνει το Συμβούλιο και τρίτον να μιλήσω για τις τεχνικές δυσκολίες, δυσκολίες χρονοδιαγράμματος και συγχρονισμού σχετικά με αυτή τη γνωμοδότηση που παρουσιάζω εδώ. Πρώτο σημείο. Η θέση της Κομισιόν. πρέπει να σας πω ότι η πρόταση της Κομισιόν αν δεχόμασταν αυτό το οποίο μας παρουσιάζει η Κομισιόν στο κεφάλαιο 1β, 1β μάλλον, τότε η Επιτροπή μας θα ήταν απόλυτα καλυμμένη. Έχει συνειδητοποιήσει η Κομισιόν ότι το πρόγραμμα των τελευταίων ετών έχει ε, ε, καταλήγει κάπου, ότι πλέον τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί λόγω του ρονταρίσματος. Βλέπουμε βέβαια ότι τα κράτη-μέλη πλέον παρουσιάζουν περισσότερα προγράμματα, ζητούν περισσότερα λεφτά για να μπορέσουν να προχωρήσουν στις πληρωνές Εμείς ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της Ευρώπης 2020 είναι η άσκηση και των περιφερειακών πολιτικών. Αυτό το οποίο μας προτείνει η Κομισιόν αντιπροσωπεύει ένα 3,4% αύξηση έναντι του προσχεδίου και στις πιστώσεις πληρωμών 8,4%. Για τις πληρωμές μιλάμε. Και εμένα μου φαίνεται ότι αυτό αντικατοπτρίζει πολύ σωστά την κατάσταση. Τι γίνεται όμως στο Συμβούλιο. Την τελευταία μια μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση την πέρασα διαπραγματευόμενος με την Πολωνική Προεδρία. Και πιστεύω ότι μπορώ να διαπιστώσω με ιδιαίτερη ε, διάβια πνεύματος του τι συμβαίνει σε επίπεδο Συμβουλίου. Τα νέα που έχουμε σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης είναι ότι το Συμβούλιο θεωρεί την περιφερειακή πολιτική ως μία από τις προτεραιότητές του αλλά αντικατοπτρίζεται σωστά στις θέσεις του. Σε ορισμένες ναι, σε ορισμένες όχι. Για τις πιστώσεις υποχρεώσεων δεν αλλάζει τίποτα. Δεν το τροποποιεί το Συμβούλιο. Συμφώνησε το Συμβούλιο με την πρόταση της Κομισιόν. Αλλά προσοχή. Εμείς αυτό δεν θα πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Διότι όσον αφορά στις πλήρωμες και για να μιλήσουμε με στρογγυλά νούμερα, ένα 300 δις μείωση προβλέπει το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του 8 0,4% σημαίνει τι. Σημαίνει ότι το κόβει το Συμβούλιο και δέχεται την αύξηση μόνο του 5%. Αυτά για τις πιστώσεις πληρωμών. Και σε αυτές τις πιστώσεις πληρωμών δεν πρόκειται να καταφέρουμε καμία ευελιξία από το Συμβούλιο. Επίσης, θεωρώ ότι δεν μπορούμε εμείς αυτό να το δεχθούμε ως τελεσμένο γεγονός. Νομίζω ότι θα ήταν απαράδεκτο η Επιτροπή μας έτσι με την πρώτη να δεχθεί αυτή την πρόταση του Συμβουλίου. Διότι τελικά στο Συμβούλιο αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού. και δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Συμβούλιο το πώς θα θα κατανεμηθούν αυτά τα κονδύλια μέσα στον προϋπολογισμό και το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ένας πόλεμος αριθμών. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι απόλυτα ρεαλιστική και έχουμε μετά την εναλλακτική λύση που κάθε χρόνο την παίζουμε ως τελευταίο χαρτί. Δηλαδή εμείς ε, δεχόμαστε τις πιστώσεις ε, ε, πληρωμών και μετά έχουμε και μια μεγαλόστομη δήλωση ως παράρτημα που λέμε ότι στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής θα δεχθούμε όλα τα απαραίτητα ποσά πιστώσεις πληρωμών. Αυτή η δήλωση εδώ και 8-10 χρόνια επισυνάπτεται. Αλλά τους ρώτησα, εσείς ξέρετε αυτά τα 8-10 χρόνια αυτή η δήλωση να χρησιμεύσε σε τίποτα. Ποτέ, τίποτα. Και πέρυσι που χρειαστήκαμε παραπάνω λεφτά για τα σχέδια της συνοχής, η δήλωση αυτή δεν ελήφθη υπόψη. Και το είπα εγώ στον Προεδρεύοντα ότι όταν υπογράφουμε κάτι, μετά τα λόγια πρέπει να γίνονται έργα. Εγώ συνεργάστηκα με την, Επιτροπή, με τη γραμματεία της Επιτροπής μας, την οποία θέλω να την ευχαριστήσω για όλη τη βοήθεια που μου έδωσε και μαζί με τη γραμματεία συντάξαμε εδώ ένα πρόχειρο όπου αρχίσαμε να αναφέρουμε κάπως την πρόταση του Συμβουλίου χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνουμε τα ποσά τα οποία έπεσαν τελευταία. Αυτό όμως συμβαίνει κάθε χρόνο βέβαια. Τώρα εσείς θα θυμάστε αυτό το back to the PDB, δηλαδή η επάνωδος στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μόνο με τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχουμε πια προσχέδιο προϋπολογισμού, έχουμε μόνο το draft budget στα αγγλικά. Εμείς για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας θα πρέπει να καταθέσουμε όλες τις δυνατές τροπολογίες που μπορούμε για να επαναφέρουμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Για το άλλο πακέτο που πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε είναι τα σχέδια πιλότη και οι, προπαρασκευαστικέ και οι προπαρασκευαστικές δράσεις. Τα pilot project και τα preparatory acts, λέει ο μιλητής. Εμείς έχουμε υποβάλει προτάσεις σχετικά, πολλές προτάσεις, αλλά μόνο μία μας ήρθε. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλα αυτά τα σχέδια πιλότους που έχουν ξεκινήσει Και τώρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πιο δύσκολο Πώς θα μπορέσουμε εγκαίρως να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία θεωρώντας ότι η επόμενη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής θα γίνει 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκτός ορίου κατάθεσης τροπολογιών 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή είναι μετά από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών. Μπορούμε να βρούμε δύο λύσεις, θα τι αναφέρω και τι δύο. Πρώτη, να χρησιμοποιήσουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, 29, 30, 31 νομίζω Αυγούστου, και μια από αυτές τις μέρες να έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για αυτές τις πιθανές τροπολογίες που θα μπορούσαμε να καταθέσουμε ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στη συνέχεια θα τις ε, εγκρίναμε. Αυτές τις προτάσεις όμως τροπολογίες θα πρέπει να τις ετοιμάσουμε τώρα πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Πρέπει να μεταφραστούν, ξέρετε ποιος είναι ο κανόνας. Γνωρίζετε ότι για τη συζήτηση στην Επιτροπή θα πρέπει να έχουμε τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες και θα πρέπει να έχουμε και quorum. Πρέπει δηλαδή να έχουμε απαρτία επαρκή για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε. Μπορεί βέβαια στην πρόταση που σας ανέφερα να μην ε, είμαι και τόσο ρεαλιστής. Και η γραμματεία υπέβαλε μια πρόταση που η πρόεδρος δεν είναι εδώ, οπότε σας τη λέω εγώ. Αν μετά από τη συζήτησή μας η Επιτροπή μας συμφωνήσει ότι θα μπορέσουμε να να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τα ποσά που έκοψε το Συμβούλιο στο αρχικό ποσό της Κομισιόν, αν το αποφασίσουμε τώρα αυτό, εγώ ως εισηγητής μπορώ να παρουσιάσω από κοινού με την Πρόεδρο αυτές τις τροπολογίες και εσείς θα μπορούσατε θεωρητικά να συμφωνήσετε σήμερα και την ουσιαστική πλέον έγκριση να την δώσετε στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου. Και στις 19 Σεπτεμβρίου δηλαδή θα εγκρίνετε το τελικό κείμενο αυτής της έκδοσης. Αν δεν κάνω λάθος, οι συντονιστές ε, συζήτησαν ε, για το θέμα. Αυτή είναι η κατάσταση κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το περιθώριο το οποίο έχουμε και περιμένω την απόφαση, τη σοφή απόφαση της Επιτροπής. Okay, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σούριαν. Κύριε Βόγαν, θέλετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτήν ε, την εξαιρετική του παρουσίαση που είχε τόσα πολλά πράγματα και μας παρουσίασε και την κατάσταση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012. Νομίζω ότι ήταν ε, μια ευρεία συμφωνία στην Επιτροπή μας ε, ότι η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχή θα έχει την ελάχιστη δυνατή αύξηση πληρωμών για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το 8,4% αύξηση όπως είπε άλλωστε και ο εισηγητής. Δυστυχώς αυτή ήταν η απάντηση από τα περισσότερα κράτη-μέλη και όπως είπε άλλωστε και και ο ε, Το Συμβούλιο τώρα λέει ότι θέλουν να μειώσουν το 8,4% ε, σε 5,2% μόνο αύξηση, που σημαίνει 1,3 δισεκατομμύρια λιγότερο από αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 700 ε, εκατομμύρια λιγότερα για ε, το ε, Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και επίσης πολύ σημαντική μείωση για τα Ταμεία Συνοχή σε σχέση με αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε αντίδραση και από, απο από κάποια κράτη-μέλη παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιφέρειες στις χώρες τους που εποφελούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα Ταμεία Συνοχής και το Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις χώρες. Φαίνεται όμως ε, ότι το ε, Συμβούλιο βλέπει τώρα ότι πολλές περιφέρειες της Ευρώπης εποφελούνται σε μεγάλο βαθμό από ε, τα ταμεία συνοχής και από, τις διαρθρωτικές, από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι στο μέλλον ε, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί μια μεγαλύτερη αύξηση. Ελπίζω λοιπόν να ακολουθηθεί αυτή η τάση και ελπίζω να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση και για το 2012 αλλά και για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα σε ε, ομιλία της Πολωνικής Προεδρίας στην Ολομέλεια το, στο Στρασβούργο ότι είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ της διαρθρωτικής πολιτικής και των ταμείων συνοχής. Έχουμε λοιπόν ένα σύμμαχο στην Πολωνική Προεδρία και μπορούμε να επιμείνουμε ε, Βέβαια το Συμβούλιο όπως αναμενόταν ε, πρότεινε ακόμη μικρότερη μείωση τουλάχιστον ε, έχουμε κάποιους συμμάχους και σε ορισμένες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην Πολωνική Προεδρία. Στις 28 Αυγούστου ε, μπορεί να ε, μπορέσουμε να επανέλθουμε με καλύτερα επίπεδα ε, πολιτικής, ε, με καλύτερα επίπεδα ε, αύξησης για τα ταμεία συνοχής και για τις διαρθρωτικές πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σουρία για την εξαιρετική περίληψη, σύνοψη για το που βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι παρόλες τις διακοιμάσεις πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην σωστή πορεία και ο κύριος Σούριαν τόνισε τη σημασία αυτής της αρχής. Επίσης πρέπει να τονίσουμε όχι μόνο έναντι των κρατών μελών αλλά και τους, τον ρόλο των πολιτών ότι το, τα κονδύλια που δαπανώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχουν πρόσθετη αξία και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα οποία γίνονται και στα κράτη-μέλη. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των πολιτών όπως ε, ε, πολλές φορές. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι ώστε να μπορέσει η περιφερειακή πολιτική σε σχέση με τα διαθροτικά κονδύλια να δράσει με τον καλύτερο τρόπο. Στη χώρα μου είμαστε παράδειγμα γι' αυτό. Όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ μας, του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγα χρόνια είμαστε στο 145% όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Αυτό οφείλεται στις ε, πολλές ε, θετικές επιπτώσεις ε, και στα διαθωτικά κανδύλια και αυτά τα μηνύματα δεν περνάνε στους πολίτες επαρκώς. Υπάρχει μια πολύ σημαντική δουλειά και πρέπει να ληφθεί υπόψη και έχουμε αμελήσει. Πρέπει τα πιο καλά προγράμματα και σχέδια να μπορούν να προχωρούν και να υποστηρίζονται. Γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξει όφελος και δεν βλέπουν την ανάγκη οι πολίτες ε, να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια όπως είχε ξεκινήσει. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, να μπορέσουμε δηλαδή να αντισταθμίσουμε αυτά τα αρνητικά στοιχεία και στο περιφερειακό επίπεδο αλλά και κάποιες αρνητικές πτυχές που υπάρχουν ε, για ε, πολιτική ιδιοτέλεια από πλευράς ε, πολλών κρατών. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και το Ατλαντικό Βήμα, το Atlantic Forum για μια νέα διατλαντική πολιτική κάτι στο οποίο έχουμε ε, αρκετά εμπλακεί και πρέπει να τονιστεί ότι αυτό θα αποδείξει την πρόσθετη αξία και το όφελος του να υπάρχει αυτή η συνεργασία, να υπάρχουν προγράμματα και σχέδια τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ε, πρόσθετη αξία για αυτές ε, τις ε, περιοχές από ότι αν το κάναμε ε, επιμέρους και ατομικά. Αυτό το μήνυμα όμως δεν περνάει όπως θα έπρεπε και είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσει να περάσει το μήνυμα όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Μία πολύ σύντομη παρατήρηση θα ήθελα να κάνω μόνο όσον αφορά τον εισηγητή και τη διαδικασία. Βρίσκω ότι έχει νόημα σίγουρα να υπάρχει συνένεση, ένα συνενετικό πλαίσιο. Κάποιες παρατηρήσεις έχουμε για τις σημειώσεις, κάτω-κάτω δηλαδή, και θα θέλαμε να συμπεριληφθούν αυτές οι ε, παρατηρήσεις ε, για τα αριθμητικά μεγέθη πρέπει να αποκατασταθούν ε, τα ποσά του προσχεδίου. Θα θέλαμε να υπάρξουν κάποιες συμπληρώσεις, διότι έχει αλλάξει κάποια πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πέρα από αυτό έχουμε και το νέο κανονισμό για τα διαθρωτικά ταμεία και πρέπει να προπαρασκευάσουμε αυτή την επόμενη φάση. Πρέπει να κάνουμε κάποια σχόλια. Έχω μεγάλη προϋπηρεσία στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάντα κάναμε τέτοιου είδους παρατηρήσεις ώστε να επαρκούν τα ε, κονδύλια. Να μπορούν για παράδειγμα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εταίροι όπως ε, τους περιγράψαμε με την προηγούμενη ανακοίνωση να συμμετέχουν οι εταίροι. Μια τέτοια τροπολογία θα συντάξουμε και θα καταθέσουμε. Δεν θα είναι νέα κονδύλια αυτά και αυτό είναι σημαντικό αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να συμφωνήσουμε για τα πιλωτικά προγράμματα. Θα πρέπει να προπαρασκευαστούμε με τις παρατηρήσεις και τις σημειώσεις να μην υπάρξουν δυσκολίες όταν θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια τα διαθωτικά ε, ταμεία. Θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις και θα, συμπεριλάβουμε, θα ε, ζητήσουμε να συμπεριληφθούν στην έκθεση από τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Κύριο Σούριαν. Θα θέλατε εσείς κύριε Σούριαν να παρέμβετε. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω διότι αναφέρθηκαν κάποια πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και θα ήθελα τώρα να αντιδράσω και να απαντήσω. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας, ευχαριστώντας όλους όσους παρενέβησαν και για το πώς τοποθετήθηκαν σε σχέση με αυτά τα θέματα. Κυρίως επειδή κανείς δεν ε, είχε αντίρρηση να μην διεξαχθεί αυτή η συνεδρίαση κατά τα τέλη Αυγούστου. Νομίζω ότι αυτό από πλευράς των συντονιστών είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσει έτσι να προαχθεί. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη όσον αφορά μας τεράστιες ευθύνες και στη μικρή συζήτηση, η μικρή διαπραγμάτευση που έκανα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου κατέστη σαφές ότι αυτή είναι τεράστια ευθύνη. Πρώτον, πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φθηνή και όχι δαπανηρή, όχι υπερβολικά δαπανηρή. 1% όλο και όλο του ΑΕΠ ε, είναι οι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον προϋπολογισμό. Πρέπει να διασφαλίζουμε όμω ότι αυτά τα κονδύλια θα χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο. Διότι στα μέσα στον τύπο μιλάνε μόνο για τα σφάλματα. Όμως τα σφάλματα είναι μεμονωμένες, από περιπτώσεις. Είναι σφάλματα, ολισθήματα, κάποια λάθη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι πορευόμαστε με τον καλύτερο τρόπο και χρησιμοποιεί η Ευρώπη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα κονδύλια που έχει στη διάθεσή της. Και σε σχέση με αυτή την κρίση θα πρέπει σιγά σιγά βήμα προς βήμα να την ξεπεράσουμε και να είναι πλέον παρελθόν. Εκείνα τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν καλά τα κονδύλια που προέρχονται για ε, που στοχεύουν στην πολιτική συνοχή, αυτές οι χώρες καταφέρνουν να ξεπεράσουν την περίοδο κρίσης με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι οι χώρες εκείνες που δεν χρησιμοποιούν τέτοια κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Η Πολωνία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Είναι ένα από τα λίγα κράτη, ελάχιστα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν υπήρξε αναχέτηση, μείωση, συρρήκνωση του ρυθμού ανάπτυξης. Όχι μόνο δεν ε, βρέθηκε στο αρνητικό, ε, δεν είχε φθήνους απορία αλλά αυξήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης και τώρα για να ολοκληρώσω και να απαντήσω θα μιλήσω αγγλικά. Ομιλώ όμω ουγγρικά ενώ συνήθως παρεμβαίνω στα αγγλικά επειδή διαβιβάζεται, μεταβιβάζεται αυτή η συνεδρίασή μα και έτσι μπορούν να, με να ακούσουν τη φωνή μου στη γλώσσα μου οι πολίτε μου στη χώρα μου. Σε σχέση με οποιαδήποτε τροπολογία ή τροποποίηση είμαι φυσικά στη διάθεσή σα. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε μια καλή λύση. Και όπω ε, αναφέρθηκε σε σχέση με την Γραμματεία. Ελπίζω ότι στις 19 Σεπτεμβρίου σε εκείνη τη συνεδρία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε τις ε, τροπολογίες. Συνεχίζει στα αγγλικά ο μιλητής. Το Σεπτέμβριο λοιπόν ακριβώς θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για το κείμενο. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά. Και όσοι ήθιστε κιόλα και να, με προφορικές τροποποιήσεις ή τροπολογίες να κάνουμε τροποποιήσεις και αλλαγέ συνενετικά όσοι ήθιστε και γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ισηγητά. Κύριε Βανίστελρο, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με διαφορετικές απόψεις, ε, αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, είναι δύσκολο πολλές φορές να μπορεί κανείς να ε, βρει ε, μια άκρη. Υπάρχει η διερμηνία, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ωραία. Όταν υπάρχει συνένεση όμως από την άλλη πλευρά και συμφωνούμε ότι τα παλαιά προτινόμενα κονδύλια του προσχεδίου θέλουμε να αποκατασταθούν σε σχέση με τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί αρχικά και τα πιλωτικά προγράμματα να μπορέσουν να υποστηριχθούν και μάλιστα ενδυναμώνοντάς τα και τονώνοντάς τα και έχουμε και πολύ θετικά παραδείγματα στην Πολωνία για παράδειγμα έχουμε όμως και αρνητικά παραδείγματα για την εκροή των κονδυλίων, την απορροφητικότητα ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν πολύ καλά. Για τέτοιου είδους προγράμματα είναι η καλύτερη οδός, η καλύτερη πορεία ώστε να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση μέσω του περιφερειακού επίπεδου στο οποίο θα παρέμβουμε και θα τονώσουμε. Αν συμφωνούμε λοιπόν εφόλων αυτών, τότε μπορούμε και μια συντετμημένη, μια επιβραχημένη διαδικασία να ακολουθήσουμε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Okay, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, αν δεν διαφωνεί κανείς, ε, θα δώσουμε την εντολή στον εισηγητή να ε, συζητήσει ούτω το θέμα της του προϋπολογισμού και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι στις 12 Ιουλίου. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι σας καλοχαιρετίζω από πλευράς μου. Έχουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και πρόκειται για την αξιολόγηση μιας μακροστρατηγικής για τις περιφέρειες, ιδιαίτερα για τον χώρο της Μεσογείου και τις μελλοντικές προοπτικές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα στον κύριο Αλφόνση, εισηγητή, να δώσω τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας πρέπει να σας πω σε όλους που ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα ότι είμαι απόλυτα ανοιχτός για να ακούσω τις γνώμες και τα σχόλια που θέλει ο καθένας να μου στείλει. Γιατί αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα πολλούς βουλευτές που προέρχονται από την περιοχή. Μια πρώτη μακροπεριφερειακή πολιτική ξεκίνησε στην Ευρώπη γύρω από την Βαλτική, μια μακροπεριφερειακή στρατηγική. Το 2009 λοιπόν και το 2011 είχαμε τον απολογισμό και λέει η Κομισιόν ότι πετύχαμε επιτυχώς αηφορία στο περιβάλλον, ενίσχυση της ευημερίας της περιοχής, προσβασιμότητα και θελκτικότητα της περιοχής, ε, ασφάλεια. Και σύμφωνα με την ίδια έκθεση της ε, Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να εμπνευσούμε από αυτό το πρόγραμμα και για μια μελλοντική πολιτική για τον Βούναβη και άλλες περιφέρειες οι οποίες έχουν ε, είτε παραλιακή είτε άλλη Η Ουγγρική Προεδρία εξέφρασε λοιπόν το ενδιαφέρον της ε, για την μακροπεριφερειακή στρατηγική για τον Δούναβη και μας κάλεσε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας για μεγάλες μελλοντικές μακροπεριφερειακές εργασίες. Βέβαια πέρα από το όχι νέες υποδομές, όχι νέες χρηματοδοτήσεις, όχι ε, νέα, νέος, ε, νέα νομοθεσία, λένε ναι σε άλλα πράγματα. Και εμεί εγκρίναμε ένα ψήφισμα της κυρίας Δανούτα Γιούμπνερ για το 2011 για μια στρατηγική για τον Ατλαντικό. Εκεί αναφερόμαστε σε συνεργασία και συντονισμό σε πολλά επίπεδα, χωρίς όμως νέα κονδύλια και θέλει αυτή η στρατηγική να ξεκινάει από τη βάση στην κορυφή ξεκινώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το κοινοβούλιο μας λοιπόν έχει ήδη αναφέρει πόσο σημαντικό είναι να επεκταθεί αυτή η πολιτική πέρα από την πρωτοβουλία του Δούναβη και τη Βαλτική. Για τις πολιτικές συνοχής ε, πρέπει να σκεφτούμε σε τι μπορούν να προσφέρουν αυτές οι πολιτικές συνοχής, πόσο μπορούμε εμείς ε, να εφαρμόσουμε νέα χρηματοπιστωτικά μέσα σαν αυτά που μας ε, δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πολιτικές συνεργασίες και καλής γυτνίασης. Και αυτό μέσα στα πλαίσια του μεσογειακού χώρου που είναι ένας χώρος σαφέστατος για την άσκηση μιας τέτοιας στρατηγικής. Έχουμε ελάχιστη διάρθρωση και δομή σε αυτή την περιοχή. Θαλάσσιες μεταφορές ε, είναι ελάχιστα ανεπτυγμένες στην μεταφορά εμπορευμάτων, ενώ θα έπρεπε να αποτελούν την καρδιά της αηφορίας για τις μεταφορές. Τα νησιά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Οι σχέσεις τους ε, είναι κυρίως με την υπηρετική χώρα, ε, χώρα του κράτους στο οποίο ανήκουν και μόνο μια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αναπτύξει τις σχέσεις. Η ποιότητα του περιβάλλοντος είναι σημαντική πρόκληση για τη Μεσόγειο που είναι κλειστή χαθάλασσα με μεγάλη βιοπικιλότητα και όπου η κίνδυνη από τις θαλάσσιες μεταφορές είναι ιδιαίτερη υψηλή. Ε, οι παραλίες όπου αυξάνεται ο πληθυσμός ε, και ο τουρισμός. Το μεσογειακό κλίμα δημιουργεί ένα περιβάλλον κοινό για όλη την, τη λεκάνη και κοινή γεωργική, και, και γεωργική παραγωγή και έχουν όλοι τον ίδιο κίνδυνο περκαγιών. Πρέπει λοιπόν επίσης να λάβουμε υπόψη την πολιτιστική κληρονομιά που είναι και ο πολιτιστικός πλούτος και ο γλωσσικός πλούτος. Μια άλλη πρόκληση για την Νότια Ευρώπη είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως η ηλιακή ενέργεια. Η πρόκληση θα μπορούσε να δραχτεί καλύτερα μέσα από ένα ενιαίο σχέδιο. Μια τέτοια στρατηγική δεν πρέπει να ξεκινήσει από την κορυφή, πρέπει να σεβαστεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και να μπορέσει να προωθήσει σχέδια με μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη άξια. Εγώ θα ήθελα δύο μακροπεριφέρειες να καλύψουν το πρόγραμμα στην Δυτική και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή η Αδριατικοϊονική περιοχή. Το χρονοδιάγραμμα που προτείνω είναι έγγραφο εργασίας ε, μέσα Οκτωβρίου 2011. Θα συζητηθεί τον Δεκέμβριο και η ψηφοφορία θα μπορούσε να γίνει σε αρχές του 2012. Μία μήνυα ακρόαση θα γίνει σε επόμενες συνεδριάσεις ε, για τις ε, μήνυ πρωτοβουλίες στην αδριατικοϊονική ζώνη. Θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ με όλους τους και οδείς από τις άλλες πολιτικές ομάδες και τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους. Ε, σας ευχαριστώ θερμά για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Πρώτος ο κύριος Τάμας Ντόιτς, παρακαλώ. στο πολύ. Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο, κυρίες και κύριοι, έχοντας ακούσει την παρουσίαση του κυρίου Αλφόνση, θα ήθελα να προσθέσω τρεις προτάσεις, τρεις σκέψεις όσα μας είπε ο κύριος Αλφόνση και που στοχεύουν ακριβώς στην κατεύθυνση των παρατηρήσεων που έκανε ο ίδιος ο κύριος Αλφόνση όπως μας τις παρουσίασε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι με την επικέντρωση αυτή στα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλφονσί με τις αρχές και τις προτάσεις που παρατηρεί για το ρυθμό που διέπει και τα στοιχεία που διέπουν την έκθεση του συμφωνώ με όλα αυτά. Με όλα αυτά. Ως κοιόδης εισηγητής του ΕΛΚΑ πρέπει να πω ότι συμφωνώ. Τώρα, Τούτου λεχθέντος. Θα ήθελα να πω ότι τρία σχόλια θα ήθελα να προσθέσω που νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο να σημειωθούν και να ληφθούν υπόψη όσον αφορά την εργασία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε την πέμπτη έκθεση για τη συνοχή. Μία έκθεση η οποία συζητήθηκε ευρέως και προκάλεσε πολλές συζητήσεις και που συμπεριλαμβάνεται και η σκέψη ότι για την προπαρασκευή και την προετοιμασία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πρώτα μία αξιολόγηση που πρέπει να γίνει. Αξιολόγηση των δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών για την περιοχή της Βαλτικής αφενός για τις περιοχές και χώρες της Βαλτικής και αφετέρου για τη στρατηγική για την λεκάνη του, Δούναβη ιδιαίτερα την Ουγγρική Προεδρία και όλα ε, που βρίσκεται υπό μορφή, υπό ε, εφαρμογή και αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Αλφόνση στην εισαγωγή του θα πρέπει να αποτελούν ένα εγγενές τμήμα, ένα οργανικό τμήμα της αξιολόγησης των σημερινών στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές στρατηγικές. Πρέπει να αποτελούν μέρος της έκθεσης λοιπόν. Δεύτερον, πρέπει να καθορίσουμε ποια είναι εκείνα τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν και καθιστούν λειτουργικές τις δύο μακροπεριφερικές στρατηγικές που ήδη υφίστανται για τη Βαλτική και τον Δούναβη. Στην πέμπτη έκθεση συνοχής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καθώς επίσης και σε όλα τα έγγραφα που αφορούν τη μελλοντική πολιτική σύνοχή που ήδη δημοσιεύθηκαν και συζητήθηκαν όλα αυτά λοιπόν τα έγγραφα στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή πρέπει να γίνει να επιτευχθεί μια ανάλυση, μια αξιολόγηση των δύο αυτών μακροπεριφερειακών στρατηγικών που προανέφερα και γι' αυτό θα ήταν λοιπόν σημαντικό η δική μας Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να καθορίσει Ποια θα είναι εκείνα τα κριτήρια που θα επιτρέπουν να γίνει αυτή η συγκριτική αξιολόγηση αυτών των αμφότερων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για την Βαλτική θάλασσα και για τον Δούναβη δηλαδή επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω αυτές τις δύο μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Και αυτό είναι το ότι αυτή η έκθεση συμπίπτει και δεν παραλλήλου με τη συζήτηση για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013 και με την εκπόνηση των μελλοντικών κανόνων και διατάξεων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική συνοχή που θα καθορίζει την πολιτική συνοχή στο μέλλον. Συζήτηση που έχει κύριο ρόλο και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σε σχέση με όλα αυτά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Είναι εκ των όνου κάνευ. Εμείς <clears throat> να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και αναμφίσιμα στις τοποθετήσεις μας και όσον αφορά τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουμε και όσον αφορά τις δυνατότητες που θα πρέπει να προσφέρουν οι μελλοντικές πολιτικές συνοχής για τις μακροπεριφερειακές πολιτικές. Και επαναλαμβάνω, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις νέες στρατηγικές μακροπεριφερειακές πολιτικές στο μέλλον, χρειάζεται συγκεκριμένη πολιτική βούληση και σθένος Ίσως όμως δεν είναι το μόνο το οποίο αφορά τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή πολιτικοί Λόγοι. Πρέπει να αναλυθούν αυτά τα πράγματα, τα πράγματα υπό ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι υπό ένα στενό πολιτικό ιδιωτελές πλαίσιο. Πρέπει να αναλύσουμε τον πιθανό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αυτές οι μακροπεριφερειακές πολιτικές καθ' όλη την περίοδο κατά την οποία θα ισχύουν και θα διαρκούν. Δηλαδή μέχρι και το 2020 και για τη ζώνη και της Μεσογείου. Είπε κάτι ο κύριος Αλφονσί το οποίο θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Και αυτό είναι το ότι θα πρέπει ίσως να υπάρχουν δύο στρατηγικές μακροπεριφερειακές όσον αφορά τη ζώνη γύρω από τη Μεσόγειο. Προσέξτε, ο αριθμός δεν είναι το σημαντικό αν θα είναι μία στρατηγική, δύο στρατηγικές. Όμως με τις διαφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα που υφίστανται και όλα αυτά συνολικά αληθεύει ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ε, θέματα. Αν όμως έχουμε μία μακροπεριφερειακή πολιτική για τη Μεσόγειο θα πρέπει να είναι μία ενιαία και μία ολοκληρωμένη πολιτική για τη Μεσόγειο και όχι δύο ή περισσότερες ξεχωριστές και κατακαιρματισμένες πολιτικές. Από την άλλη τώρα πλευρά, ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι εδώ σε αυτή την έκθεση πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι αυτή θα είναι η κύρια πιθανότητα να είναι η τρίτη δηλαδή στρατηγική μακροπεριφερική μετά τον Δούναβη και τη Βαλτική ακριβώς η Μεσόγειος και η, όπως λέει ο κύριος Αλφονσί θα πρέπει να καθορίσουμε σαφώς τη θέση μας. Θα είναι η τρίτη αυτή η μακροπεριφερική πολιτική ή θα υπάρχει και τέταρτη σε συντονισμό με τις υφιστάμενες δύο. Λοιπόν, Συνοψίζω, πρέπει να καθορίσουμε βασικά θεμελιώδη κριτήρια για την υλοποίηση της στρατηγικής για τη Βαλτική και το Δούναβη. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις πολιτικές πέρα από το στενό πλαίσιο του 2013 σε ένα ευρύτερο χρονορίζοντα και για την πιθανή μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Μεσόγειο να αποφασίσουμε είναι καλύτερο να υπάρχει μία τέτοια ενιαία πολιτική ή δύο ξεχωριστές σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Και η συνάδελφος Λουκατσεύσκα έχει τον λόγο τώρα παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εγώ συμφωνώ, είμαι υπέρμαχος ε, των μακροπεριφερειών γιατί πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους ε, για την καλύτερη προστασία των φυσικών πόρων, ε, της χρήσης και εκμετάλλευσής τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επίσης της αξιοποίησης του τουριστικού δυναμικού, όπως επίσης και του ανθρώπινου δυναμικού των περιφερειών αυτών. Επίσης, Μπορούμε έτσι να εκμεταλλευτούμε καλύτερο συντονισμό όταν πρόκειται για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως, ζήτησα το λόγο γιατί ο κύριος Αλφονσί στα εισαγωγικά του σχόλια φάνηκε να έλεγε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ε, για το Δούναβι, ε, για την ε, Βαλτική θάλασσα και ότι μπορούμε να βασιστούμε στο παράδειγμα αυτών των δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών για να το εφαρμόσουμε και σε άλλες ε, περιφέρειες. Για παράδειγμα, η περιοχή των Καρπαθίων, επειδή γνωρίζω πολύ καλά και το δυναμικό της περιοχής αυτής, αλλά και των ε, εξαιρετικών πόρων της, ήθελα να ρωτήσω αν θα, υπάρξουν, αν θα υπάρξει ιδιαίτερη ε, προσοχή και για την περιοχή αυτή. Φαντάζομαι ότι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να έχουν άλλες ευαισθησίες. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν θα υπάρξει κάποια στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων ε, στο άμεσο μέλλον ή αν θα επικεντρωθούμε μόνο σε αυτές ε, ε, τις μακροπεριφέρειες, στις μακροπεριφέρειες τι οποίες ανέφερε ο κύριος Αλφονσί. Γιατί όταν υπάρχει μια περιφέρεια με ενδιαφέρον δυναμικό, όπως η δική μου περιφέρεια, πιστεύω ότι θα έπρεπε να της δίνεται μια ευκαιρία, αν κάνουμε αυτή την προσπάθεια, για άλλες περιφέρειες οι περιφέρειες που θέλουν να είναι δυναμικές από πλευράς διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει και εκείνες να έχουν μια ευκαιρία για να μπορέσουν να αποτελέσουν μακροπεριφέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω μια απάντηση. Θα υπάρξει δυνατότητα μακροπεριφέρειες στην περιοχή των Καρπαθίων. Αν η ομορφιά των περιφερειών ήταν κριτήριο επιλογής, τότε η περιοχή των Καρπαθίων σίγουρα θα επελέγεται. Είμαι στεναρά πεισμένος γι' αυτό. Κύριε Σαροκάτση παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σαγκουράκης. Ε, Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν νομίζω ότι η μακροπεριφέρεια της Μεσογείου, αν και κάποτε γίνει, θα είναι σημαντικά διαφορετική από, από αυτή του Δούναβη και της Βαλτικής, για τον πολύ απλό λόγο ότι συνορεύει με τη Βόρεια Αφρική και φυσικά οι χώρες αυτής της περιοχής έχουν άλλα προβλήματα, άλλα ζητήματα από αυτά που έχει η Κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο κιόλα ίσω δεν είναι και τόσο χρήσιμο να γίνονται συγκρίσει ε, όπω επιχειρήθηκε. Το δεύτερο, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και από τον εισηγητή υπήρχε έτσι, ε, είχα την αίσθηση ότι ε, απέφυγε να αναφερθεί και σε ορισμένα άλλα κοινά ζητήματα στη Μεσόγειο, τα οποία όμως αν δεν αντιμετωπιστούν δεν θα μπορεί να γίνει λόγος πραγματικά για μια μακροπεριφέρεια. Και ενώ καταρχήν εάν θα υπάρχει ένα πνεύμα που να ενισχύει τη συνεργασία, την ισότιμη συνεργασία των χωρών και των λαών της περιοχής ή αντιθέτως ε, θα υπάρχει ένα πνεύμα ανταγωνισμού ή ανταγωνιστικότητας. Και αναφέρομαι στο εξής συγκεκριμένο πράγμα. Ένα πρώτο ζήτημα που είναι κοινό επίσης στην ε, Μεσόγειο είναι η αντισυσμική προστασία. Δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο από τον εισηγητή. Ένα δεύτερο ζήτημα που είναι επίσης κοινό και ειδικά σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης όπως βιώνουμε τώρα είναι ακριβώς τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα του ευρωπαϊκού νότου τα οποία συζητούνται ευρέως. Εάν τα προβλήματα αυτά που είναι προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης δεν αντιμετωπιστούν σε μια ισότιμη βάση τότε δεν μπορεί να υπάρξει κατά τη γνώμη μου, μια ε, μακροοικονομική ε, περιφέρεια στην ε, Νότιο Μεσόγειο. Ένα από τα ζητήματα αυτά είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός θα εξοκολουθεί να είναι ένα στοιχείο ανταγωνισμού ποιος έχει το φτηνότερο εργατικό κόστος ώστε να τραβάει τους περισσότερους τουρίστες ή θα γίνει σε άλλη βάση. Και ποια θα είναι αυτή η βάση. Δεύτερο ζήτημα είναι η κρίση στην, στα ναυπηγεία Μεσογείου. Θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική ας πούμε να παράγει χιλιάδες ανέργους ή θα πρέπει να αλλάξει μια πολιτική σε ισότιμη συνεργασία ε, στην ε, Μεσόγειο. Και ένα τρίτο ζήτημα βεβαίως αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Αυτά είναι ζητήματα που δεν, ε, δεν απασχόλησαν τον εισηγητή. Καταλαβαίνω ότι το κάνει, γιατί όσο είναι το καπιταλιστικό σύστημα, <laughs> πολύ δύσκολο θα υπάρχει μια ισότιμη συνεργασία, αλλά τότε πρέπει να είμαστε και πιο ε, ειλικρινεί και να ξέρουμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για αυτή σας ε, την παρατήρηση. Κορώνα παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι ο συνάδελφος Αλφονσί είπε έστω και γενικώ, υπέδειξε μάλλον έστω και γενικώ, τη γενική τοποθέτηση της έκθεσής του για ένα θέμα τόσο σημαντικό όπως είναι αυτό των μακροπεριφερειών. Εγώ θα είμαι και όδης εισηγητής εκ μέρους σοσιαλιστικής ομάδας για αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό όπως υπόθηκε και πριν να έχουμε μία αξιολόγηση συγκεκριμένη αξιολόγηση για το πώς. Λειτουργήσε το πρώτο πείραμα για τις μακροπεριφέρειες στη Βαλτική και στο Δούναβι. Πρέπει να έχουμε μία συγκεκριμένη αξιολόγηση για το θέμα αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω αφορά στο γεγονός ότι το μέσο των μακροπεριφερειών είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις και ένα ιδιαίτερα έντονο και ισχυρό σχέδιο. Φτάνει όμως οι στόχοι να είναι λίγοι, συγκεκριμένοι και σε θέση να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η συμβουλή μου θα ήταν κατά συνέπεια να αποφύγουμε στην οικοδόμηση του σχεδίου των μακροπεριφερειών να πούμε, να αναφέρουμε πολλές, πολλούς και γενικούς στόχους. Χρειάζεται μία αυστηρή διατύπωση του στόχου που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Φυσικά έχω την πρόθεση να συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους συναδέλφους για να έχω ένα θετικό αποτέλεσμα με αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βλάσακ παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Και εγώ εκτίμης, εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι συζητούμε αυτό το θέμα. Γιατί αν δει κανεί την έκθεση και μάλιστα την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τις σημερινές πρακτικές αλλά και τις μελλοντικέ προοπτικές. Και όταν κάνουμε λόγο για τη Μεσόγειο, ως ένα σύνολο σφαιρικά, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε την πείρα την εμπειρία που έχουμε όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ μεσογειακών χωρών όπως ε, για παράδειγμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή την ε, Ένωση Δήμων και Περιφερειών. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα καλής συνεργασίας, ήδη υπάρχουν κάποια αποτελέσματα από πρώτο χέρι. Ας δούμε λοιπόν, ας αξιολογήσουμε πώς επετεύχθη αυτή η συνεργασία, πώς επετεύχθησαν αυτά τα αποτελέσματα και ίσως αυτά μπορέσουν να εμπνεύσουν, να μας εμπνεύσουν για το έργο μας, την εργασία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ' αυτών. Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι κάθε χώρα μπορεί να θεωρείται ως ένα τμήμα, ένα μέρος μιας μακροπεριφέρειας. Ο συνάδελφος ανέφερε την περιοχή των Καρπαθίων θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στις Άλπεις παράδειγμα και επίσης και στην Ευρώπη ως ένα ευρύτερο σύνολο. Διερωτώ με, αυτή είναι η σωστότερη προσέγγιση σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική. Μια τέτοια προσέγγιση. Το εκτιμώ λοιπόν ότι θα έχουμε μια έκθεση από ε, αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να αναθεωρήσουμε, να επαναξιολογήσουμε αυτές τις μακροπεριφερειακές πολιτικές όπως για την πολιτική για την Βαλτική που ξεκίνησε υπό την Σουηδική Προεδρία και να αναθεωρήσουμε και να δούμε, να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, μακροπεριφερειακής πολιτικής για τον Δούναβη και να δούμε τι μπορούμε να συναγάγουμε ως συμπεράσματα. Ένα ερώτημα. Η Ευρώπη συνολικά είναι μια μακροπεριφέρεια. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Η κυρία Σάντσια Σμιτ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλφονσί όταν ξεκίνησε να μιλάει για τους ε, στόχους ε, της μακροπεριφέρειας του Δούναβη, ε, σίγουρα πρέπει να συμφωνήσουμε για το ποιοι είναι οι στόχοι μιας μακροπεριφέρειας και ποιοι οι γενικοί στόχοι. Δεν νομίζω ότι προορισμός της Ευρώπης είναι να καλυφθεί από μακροπεριφέρειες. Οι μακροπεριφέρειες έχουν ένα συντονιστικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές και στη λεκάνη της Μεσογείου εμείς έχουμε πολλές πολιτικές οι οποίες επικαλύπτονται πέρα από την περιφερειακή πολιτική της πολιτικής συνοχής έχουμε και την πολιτική της. και νομίζω ότι αυτή η δράση των μακροπεριφερειών θα πρέπει να έχει περιορισμένους ε, στόχους αναφέρθηκαν στην παρουσίαση σίγουρα το περιβάλλον είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Οι μεταφορές επίσης. Εμείς ε, έχουμε στρατηγικές οι οποίες ε, ε, που, πολιτικές που μπορούν να, να είναι απόρρια και των στρατηγικών για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μακροπεριφέρεια με μακροπεριφέρεια. Δεν είναι συνταγή που εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της Ένωσης κατά τον ίδιο τρόπο. Ε, σας, ε, τι σας κινεί να ε, τίνετε προς ε, το διαχωρισμό των δύο μακροπεριφερειών στη Μεσόγειο, τη Δυτική και την Ανατολική. Τι σας οδηγεί σε αυτό. Okay, dann Mr. Kelly. Εντάξει, ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ εσάς για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η συζήτηση για τις μακροπεριφέρειες αποκτά ρυθμό και επιταχύνεται. Έχουμε την Βαλτική και το Δούναβη και συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση των όσων έχουν γίνει προτού συνεχίσουμε αυτή την πορεία και προχωρήσουμε. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και η παρατήρηση που έγινε από τον κύριο Καρόζο νομίζω είναι σωστή η παρατήρηση. Πρέπει να υπάρχει πρόσθετη αξία που θα δημιουργείται και να υπάρχουν εξειδικευμένοι στόχοι, χειροπιαστοί στόχοι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τον Ατλαντικό, για την Ατλαντική περιφέρεια, ο θαλάσσιος τουρισμός, τα θαλάσσια αθλήματα και ιδιαίτερα η αιωλική ενέργεια καθώς και η ε, εκμετάλλευση αυτής της πτυχής μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία και σίγουρα μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί και μέσω των, ε, της παλήριας ε, και των, της ε, πλημμυρίδας και της άμποτης να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λοιπόν με ένα συντονισμένο τρόπο μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη αξία σε συγκεκριμένα χειροπιαστά προγράμματα και να δώσουν ωφέλη. Και τότε φυσικά κάτι θα μπορεί να γίνει δεν μπορεί να είναι επί παντός του επιστητού και επί ε, εφόλων των στόχων. Πρέπει να είμαστε πολύ στοχοθετημένοι και εξειδικευμένοι και έτσι να έχουμε αξιολογώντας τα όσα έχουμε πετύχει να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και για άλλες περιφέρειες. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. Σον θα με απογοήτευε αν τώρα το θέμα των αθλημάτων δεν αναφερόταν, αλλά αναφέρθηκε εξαιρετικά. Επόμενος, ο κύριος Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, και εγώ ευχαρίστω να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για τις περιφέρειες σε όλα τα μεγέθη και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Σπούδασα γεωγραφία στο παρελθόν και ένα πράγμα κατανόησα ότι δεν είναι πάντα σαφές και δεδομένο το τι είναι κάποια περιφέρεια και μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η Ευρώπη. Και η Ευρώπη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ευρύτερη περιφέρεια. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο ε, όπου μπορούμε να είμαστε οι πιο αποτελεσματικοί. Το να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες, ε, στο επιχειρήν, αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Δεν είναι μόνο ο προσδιορισμός μιας περιφέρειας αφεαυτής, δεν θα πρέπει λοιπόν να διασπαθίζουμε τα κονδύλια και το δυναμικό μας. Δεν πρέπει να αντλεί κανείς ε, το δυναμικό από εκεί στο οποίο ανήκει, δηλαδή το τοπικό επίπεδο. Και βλέπουμε ότι η μακροπεριφέρεια και η συνεργασία στις μακροπεριφέρειες είναι η συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Και όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν για παράδειγμα να χορέψουν έναν χορό όπως μια Πολο... Ε, Πολωνέζα της Πολωνίας αν δεν υπάρχει συντονισμός δεν μπορεί να χορέψει κανείς κάποια πράγματα πρέπει να αποσαφινιστούν πρέπει να καταστεί σαφές πού έγκυται η πρόσθετη αξία των μακροπεριφερειών Μπορεί να είναι ωραία μια περιφέρεια, εξαιρετική ομορφιάς, με εξαιρετικά τοπία, η μουσική, αλλά αυτό δεν δημιουργεί αφ' αυτού πρόσθετη αξία. Πρέπει να διαρωτηθούμε τι προσφέρει η μία μακροπεριφερειακή τέτοια προσέγγιση και ποια είναι η πρόσθετη αξία που προσφέρει. Τα κονδύλια προέρχονται ούτως ή άλλως από τα κράτη-μέλη και με άλλους τρόπους θα αντλούνται και θα χρησιμοποιούνται στις, από τις περιφέρειες. Εξαρτάται λοιπόν το τι εννοούμε και περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για τα σωστά κριτήρια που πρέπει να επιλέγονται και γι' αυτό μια συζήτηση επ' αυτών των θεμάτων είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Είναι θετικό να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση που θα είναι σημαντική για την Ευρώπη και για το χώρο της Μεσογείου φυσικά ιδιαίτερα σημαντικό αυτό μόνο που δεν θέλω ένα πράγμα δεν θέλω οι μακροπεριφέρειες να αποτελέσουν ένα ψεύδο επιχείρημα, ένα προσχηματικό επιχείρημα για τα κράτη-μέλη για να πούν «Α, δεν χρειαζόμαστε πια περιφερειακή πολιτική εφόσον έχουμε καταφέρει σε αυτό το επίπεδο να δράσουμε». Η πρόσθετη αξία προέρχεται από τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών. Και βλέπετε ότι οδηγούμαστε προσχηματικά σε μια επανεθνικοποίηση των πολιτικών μας υπό το πρόσχημα της, των μακροπεριφερειών. Παράδειγμα, Ατλαντική μακροπεριφέρεια. Μπορεί κανείς να φανταστεί πολλά πράγματα. Μακροπρόθεσμα όμως η περιφερειακή πολιτική ε, αποτελεί, θα έλεγα, ε, ε, παρακάμπτεται. Παρακάμπτεται επειδή κάποιοι θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνει και ιδιωτελώς να δράσουν. Όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να δούμε με ποιους μηχανισμούς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα πράγματα και να τα οδηγήσουμε προς τους σωστούς προσανατολισμούς. Αν έχουμε λύσεις για τα, για λιμάνια, ε, για το ένα ή το άλλο, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε μια τέτοια πολιτική να εξυπηρετήσει στόχους επί του επιστητού. Γι' αυτό λοιπόν η εθνική πολιτική δεν πρέπει να παρακάμπτει την περιφερειακή πολιτική. Χρειαζόμαστε τις σωστές απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω τον λόγο για να ολοκληρώσει ο εισηγητής. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει να μας πει κάτι. Είναι κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόν και μπορεί να παρέμβει. Παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Κάτρι Ούσταλ, σύμβουλος ε, στον Γενικό Διευθυντή ε, της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είμαι καινούρια στο συγκεκριμένο ε, τμήμα, αλλά έχω ασχοληθεί με την περιφερειακή ανάπτυξη και στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ε, έκθεση αυτή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ολοκληρώσει την κατάρτιση της στρατηγικής για το Δούναβι η οποία δρομολογήθηκε τώρα στην Λόγο περιφέρεια και τώρα προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα και στην περιφέρεια της Βαλτικής αλλά και στην περιφέρεια ε, του, του Δουνάβεως ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι συμμετέχοντες να μπορούν να ε, είναι βέβαιοι για τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής. Όσον αφορά τώρα το μέλλον των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόλις άρχισε την, τον προβληματισμό της πέρα από τις δύο υπάρχουσες ε, στρατηγικές, ε, το 2013 θα υπάρξει μία αναθεώρηση ε, ολόκληρη της προστιθέμενης αξίας των δύο μικροπεριφερειακών στρατηγικών, μακροπεριφερειακών στρατηγικών που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε για την ώρα είναι ότι είναι μάλλον νωρίς για να αξιολογήσουμε ε, τα αποτελέσματα μια τέτοια στρατηγικής. Δεν αφορά μόνο την κατάρτιση ενός εγγράφου. Το θέμα είναι αν οι στόχοι ε, εκπληρώνονται. Μερικές μόνο ιδέες μπορώ εγώ να παραθέσω, ότι τις οποίες μπορείτε ενδεχομένως να συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας, ε, που μας ενδιαφέρει βέβαια πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς ε, στην έκθεση για τη Βαλτική, ε, την οποία λάβαμε πριν από μερικές εβδομάδες και δείχνει τα αποτελέσματα της στρατηγικής για τη Βαλτική μέχρι τώρα. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω είναι τα εξή. και κάποια μάλιστα αναφέρθηκαν ήδη στην συζήτηση σήμερα. Ο ρόλος και η ευθύνη των ε, συμμετεχόντων. Και το, ο βαθμός της δουλειάς ε, που σημαίνει κάτι τέτοιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Ενδεχομένως να υπάρξει, να υπάρξει η παρεξήγηση ότι αν ζητήσουμε κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει, θα το κάνει και έτσι θα έχουμε μια πολύ ωραία μακροπεριφερειακή στρατηγική. Δεν πρόκειται να δουλέψει κάτι τέτοιο. Και από τη Βαλτική και από το Δούναβη είδαμε ότι χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης και από τα κράτη-μέλη και από τις περιφέρειες και για όλους τους ε, φορείς που συμμετέχουν επιτόπου στις περιφέρειες. Χωρίς αυτούς δεν μπορούν καν ε, να ε, σταθούν οι στρατηγικές αυτές, ε, πολλό δε μάλλον να αποδώσουν αποτελέσματα. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα της στρατηγικής για το Δούναβι, αλλά πρέπει να παραμείνει αυτό το υψηλό επίπεδο ακόμη και μετά από την κατάρτιση του εγγράφου στρατηγικής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η στρατηγική ολοκληρωθεί ως έγγραφο, τότε τα εθνικά σημεία επαφής, ε, οι συντονιστές των τομέων προτεραιότητας πρέπει να τοποθετήσουν το θέμα αυτό ως αρχική τους προτεραιότητα προτεραιότητα και να δουλεύουν για το θέμα αυτό επί καθημερινής Διαφορετικά δεν μπορεί να τους υποκαταστήσει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα επίπεδο ε, δέσμευση όχι μόνο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από όλου όσου συμμετέχουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν υπάρξει μια στρατηγική στο πλαίσιο της οποίας ε, ένας ε, σημαντικός αριθμός ε, χωρών που συμμετέχουν δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να δούμε την, τις δυνατότητες που υπάρχουν ε, για συμμετοχή των χωρών αυτών σε ισότιμη βάση, γιατί πρέπει να υπάρχουν ε, προφανώς ε, να υπάρχει ίση δέσμευση από όλους τους συμμετέχοντες και να είναι και ίσα τα ωφέλη για όλους. Νομίζω επίσης αναφέρθηκε και στη συζήτηση σήμερα το γεγονός ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μεταξύ τους οι στρατηγικές. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία ε, θεωρούμε ότι είναι ε, χρήσιμα σε αυτή τη συζήτηση. Για παράδειγμα, κάθε στρατηγική θα έπρεπε να έχει το μικρότερο ε, δυνατό αριθμό στόχων πρέπει να είναι απολύτως σχετικές με την περιφέρεια για την οποία καταρτίζεται η εν λόγω στρατηγική. Νομίζω ότι θα ολοκληρώσω εδώ. Περιμένουμε εναγωνίως ε, την έκθεση και ειδικότερα τα κριτήρια που θα μας επιτρέψουν να προσμετρήσουμε την προστιθέμενη αξία και στα οποία βέβαια θα βασιστούμε στα επόμενα δύο χρόνια πριν από την αξιολόγησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής τώρα θα λάβει τον λόγο για να ολοκληρώσει. Ο κύριος Αλφονζή παρακαλώ. Euh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις τους. Βρισκόμαστε στην αρχή της δουλειάς μας, επομένως σύν χρόνο πιστεύω ότι θα προοδεύσουμε και θα καταλήξουμε σε απαντήσεις ε, που θα μπορέσουμε από κοινού ε, να ε, ε, απαντήσουμε. Ακούσαμε ότι, για παράδειγμα, ότι είναι καλή χρονική στιγμή της έκθεσης και άλλοι συμφώνησαν ότι τώρα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε με το θέμα της, των μακροπεριφερειών γιατί έχουμε αρκετή εμπειρία, είμαστε σε φάση προγραμματισμού για τις περιφερειακές πολιτικές. Τώρα λοιπόν πρέπει να προβληματιστούμε, να αναρωτηθούμε πώς, ε, πώς οι, οι μακροπεριφερειακές αυτές στρατηγικές ε, με την εμπειρία των παραδειγμάτων του Δουνάβεως και της Βαλτικής πώς είναι δυνατόν λοιπόν να είναι μια τέτοια στρατηγική ανοιχτή σε όλες τις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης που το επιθυμούν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, είναι μια προσπάθεια η οποία έχει νόημα μόνο αν υπάρχει βούληση για συνεργασία ε, αυθορμήτως ε, των περιφερειών αυτών. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλει κανείς μια στρατηγική και να περιμένει να έχει αποτελέσματα. Κοιτάξτε, η κυρία Χιουμπνερή η πρόεδρός μας, ε, είχε προγραμματίσει μία ακρόαση με τις ε, περιφέρειες Αδριατικής και του Ιουνίου που ε, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για μια τέτοιου είδους στρατηγική. Είναι ανοιχτό λοιπόν το ζήτημα. Είναι προφανές ότι θα το συζητήσουμε, ότι θα καταλήξουμε από κοινού σε συμπεράσματα. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν σε αυτήν την τεράστια μεσογειακή περιφέρεια να υπάρξουν ε, μακροπεριφέρειες ε, είναι κάτι το οποίο θα προκύψει αυτή τη στιγμή θα εκφραστεί η βούληση από τους συμμετέχοντες στη στρατηγική αυτή. Για τον κύριο Αγκουράκη θα ήθελα να απαντήσω ότι ναι, βεβαίως χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα, χρειάζεται μια ε, οικονομική αύξηση, αλλά για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρξει μια τέτοια μακροπεριφερειακή στρατηγική, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο κλίμα στις συνεργασίες που θα υπάρξουν και για να υπάρξει και η συγκεκριμένη οικονομική ανάπτυξη. Γιατί υπάρχει ανάπτυξη που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τουριστική ανάπτυξη και υπάρχει επίσης ε, ε, μία στρατηγική που δίνει τη δυνατότητα για παράδειγμα, ε, τα ναυπηγεία να μην εγκαταληφθούν. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το ένα πρέπει να είναι εναντίον του άλλου. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τεθούν ορισμένα ζητήματα σε πολύ πιο ευρία ε, βάση. Συγγνώμη. Όσον αφορά το στόχο της συγκεκριμένης έκθεσης, ε, είναι φιλόδοξο και είναι η ύπαρξη κριτηρίων. Πρέπει να ορίσουμε κάποια κριτήρια, να πούμε ιδού η συγκεκριμένη τομής, ιδού η αξιολόγηση που κάνουμε και για ποιο λόγο μια μακροπεριφερειακή στρατηγική θα μπορούσε ή όχι να ε, έχει κάποιο νόημα σε ένα ε, τοπικό πλαίσιο. Για ε, πολλούς ε, στόχους συμφωνούμε ότι βεβαίως χρειάζονται ε, ισχυρές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βέβαια μπορεί στη συνέχεια να συνδυαστούν με, διάφορου, με διαφόρων ειδών εφαρμογές όμως πρέπει ε, δεν αρκεί ας πούμε κάποιος επειδή ζει σε μια περιφέρεια που έχει κάποιες, κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά με μια περιφέρεια που είναι τμήμα μακροπεριφέρειας ότι αρκεί κάτι τέτοιο ως κριτήριο για να υπάρξει μακροπεριφέρεια και για αυτές τις περιφέρειες ε, πρέπει να γίνει μια πολύ καλή και λεπτομερής ανάλυση και θα ήθελα επίσης να πω προς τον κύριο Φανίστελ Ρόι ότι εντάξει, σε γενικέ γραμμέ δίκιο έχει. Υπάρχει ένα κίνδυνο ε, να φτάσουμε και πάλι σε μια επανεθνικοποίηση τη περιφερειακή πολιτική. Όμω, αν οι περιφερειακές πολιτικές δεν ε, εκφράζουν την συνεργασία τους ε, με μια άλλη περιφέρεια και αρχίζουμε να μιλάμε για την προστιθέμενη αξία ε, ορισμένων στρατηγικών, τότε μπορεί πάλι να φτάσουμε σε μια επανεθνικοποίηση γιατί δεν θα υπάρξει πλέον συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και πάση περιπτώσει θα έχουμε μια στρατηγική η οποία δεν θα ταποκρίνεται σε ορισμένες προκλήσεις και η οποία θα αφορά μόνο τη Σαρδινία, την Κορσική, εν πάση περιπτώσει διάφορες περιφέρειες και όχι μια ευρύτερη ε, ε, μακροπεριφέρεια. Ε, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο τρόπος να αποφύγουμε την επανεθνικοποίηση είναι ακριβώς οι τοπικοί φορείς να υλοποιούν τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Αυτά ήταν τα λίγα σημεία που θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτή τη φάση. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα δουλέψουμε, ελπίζω αρκετά σύντομα και θα έχουμε τη δυνατότητα ε, συνεργασίας ε, με τους εκπροσώπους ε, της ζώνης Αδριατικής Ιωνίου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους για το θέμα αυτό. Ο κύριος Πίπερ, σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Σίγητα και προτείνω τώρα να διακόψουμε για λίγα λεπτά τη συνεδρίασή μας μέχρι ότου ο υφυπουργός, ο Ούγγρος υφυπουργός θα προσέλθει. Βρίσκεται ήδη εδώ. Ε, εντάξει, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εγώ βλέπω στην ίδια ψηφοφορία να περνάμε τι εκθέσει σε βέβαια, είναι πολλά Λοιπόν, μετά ξαναρχεί Αλλά σίγουρα είναι έτσι. Σε μια εκθέση είναι Δύο το πολύ. Ποιο δύο το πολύ, παιδί μου. θα ορίζει αλλά πέραν του εδώ, άντα σε έπαιρνα και ήθελε κάτι άλλο για την εξασφάλιση της Ουαλίας. Παίρνει στο Ιρλανδό και χωρίς να σου φύγει ένα ζώμα. Αυτό μόνο είδα. πάντων, δεν είναι να βγάλω ποτέ Δηλαδή, τι σχέση έχει. So, και κύριοι, Κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας τώρα και σας παρακαλώ οι συζητήσεις σας να σταματήσουν τώρα. Αγαπητοί φίλοι του ΕΛΚ ιδιαίτερα, Κύριε Τεσέρα, κύριε Φανίστερ Ρόι, κύριε Τόιρα, εσείς του ΕΡΚ σταματήστε τις συζητήσεις σας. Πολύ καλά λοιπόν, ακριβώς. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχουμε σήμερα έναν εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου για να συζητήσουμε για θέματα διαθροτικής πολιτικής. Ο κύριος Υφυπουργό ε, Κόβατς είναι παρόν και του δίνω αμέσω τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο κύριε Υφυπουργέ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ιδιαίτερη χαρά είναι για μένα να βρίσκομαι εδώ εξ ονόματος του κυρίου Τόμας Φέλεγγη Υπουργού. Και είναι η τρίτη φορά για την παρουσία της ε, Ουγγρικής Προεδρίας και της κυβέρνησής μας ενώπιον της Επιτροπή Ήτρε. Με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και μέσα στο πλαίσιο της φιλικής προς το Ευρωκοινοβούλιο Ουγγρικής Προεδρίας νομίζω καταφέραμε να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας και ως κράτος μέλος να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προεδρία και θέλουμε να συνεχίσουμε τηρώντας τι δεσμεύσεις μας έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα έναντι εκείνων των κοινοβουλευτικών επιτροπών που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα χαρτοφυλάκια του δικού μας ε, Υπουργείου, για την πολιτική συνοχή και την πολιτική ε, ανάπτυξης, ε, περιφερικής ανάπτυξης. Έχετε νομίζω πάρει την περίληψη, το hard copy της παρουσίασης των πεπραγμένων της Ουγγρικής Προεδρίας και εγώ και οι συναδελφοί μου είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας όσον αφορά τα θέματα αυτού του εγγράφου και από πλευρά τη εξάμεινη προεδρία μα είμαστε στη διάθεσή σα. Θα περάσω και θα χρησιμοποιήσω την ουγγρική γλώσσα τώρα στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε Καλησπέρα σας. Στους παρόντες αλλά και στους όσους παρακολουθούν τη συνεδρίαση μέσω του διαδικτύου. Ολοκληρώθηκε η Ουγγρική Προεδρία. Έχουμε έξι μήνες γεμάτους ε, επιτυχίες και γεγονότα. Δύο φορές ήδη ήρθα εδώ συνοδεύοντας τον Υπουργό, τώρα είναι η τρίτη φορά χωρίς Υπουργό και θέλω να σας πληροφορήσω για τις εργασίες της Ουγγρικής Προεδρίας, για την περιφερειακή πολιτική, αλλά και για το τι κάναμε μέχρι τώρα και για τις προπτικές, για τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Είχαμε μια Είχαμε μια ποικιλία πράξεων και προγραμμάτων επί Ουγγρικής Προεδρίας και η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Προεδρία μας. Μία Ευρώπη πιο ανεπτυγμένη δημιουργεί απασχόληση, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας τις ανισότητες των περιφερειών, με την Ευρώπη και στο διεθνές επίπεδο. Θέλαμε λοιπόν μια πολιτική συνοχής ισχυρή που θα μπορούσε να απαντήσει στις νέες προκλήσεις και θα μπορούσε να προωθήσει τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κατάσταση μετά την κρίση, διότι όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το maximum τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών με τα λιγότερο δυνατά κονδύλια. Και αυτό διαπιστώθηκε όπως και με όλες τις πολιτικές της Ένωσης ότι χρειάζεται ακόμα πολύ για να προχωρήσουμε. Κατά την Ουγγρική Προεδρία θελήσαμε να έχουμε προοπτικές Θέλησαμε να έχουμε ανοιχτές προοπτικές για την περιφερειακή πολιτική και θέσαμε ω στόχο την αξιολόγηση της σημασίας, της αποτελεσματικότητας και τα αποτελέσματα της περιφερειακής πολιτικής και είδαμε ή προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε και την ορατότητα. Η Ουγγρική Προεδρία έθεσε ως βασικότατη στόχο την πολιτική συνοχή, πρόβαλε και στα ΜΜΕ και σε όλους τους πολιτικούς κύκλους θελήσαμε να έχουμε μία προεδρία φιλική και συνεργατική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεργαστήκαμε στενά και με την Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να βλύνουμε τις διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία της συνθήκης της Λισαβόνας και να προχωρήσουμε από κοινού. Εμείς μιλήσαμε για τη σημασία των χωροταξικών στόχων και τη σημασία του στη στρατηγική 2020. Σε σχέση με όλα αυτά, αναλάβαμε μέτρα για τη χωροταξική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Και την πολιτική συνοχή στέλνουμε στα συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσπαθήσουμε να περάσουμε από τις αντιλήψεις πλέον, από τις ιδέες στην, στην πράξη για να εφαρμόσουμε τους νέους κανονισμούς και ρυθμίσεις και να ξεκινήσει η νέα περίοδος προγραμματισμού. Επίσης η Ουγγρική Προεδρία τόνισε διάφορες θεματικές και την ανάλυση στα διάφορα, τις ανάλυσης στα διάφορα φόρα. Ας πούμε στρατηγικός προγραμματισμός, θεματική συγκέντρωση, ολοκληρωμένη εστίαση και πολιτικές που θα προσανατολίζονται προς τα αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα σε σχέση με τα διάφορα διαμειφθέντα κατά την Ουγγρική Προεδρία να σας αναφέρω λεπτομερέστατα ποια ήταν τα αποτελέσματα. Πρώτο ήταν η προετοιμασία και έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να εγκρίνουμε ένα πολιτικό έγγραφο τέτοιου υψηλού επίπεδου για το μέλλον της, Ένωσης, της πολιτικής συνοχής στην Ένωση. Και στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Ιανουαρίου πέρασε αυτό το θέμα. Επίσης, διαπιστώσαμε ποια σημεία έχουν συνένεση μεταξύ των κρατών μελών και ποια σημεία χρειάζονται ακόμη περισσότερη συζήτηση για τις προετοιμασίες των μελλοντικών εργασιών του Συμβουλίου. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι η πολιτική συνοχή αποτελεί έναν από τους πυλώνες της, οικονομικής, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κατά συνέπεια πρέπει να τον ισχύσουμε. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων οι Υπουργοί επίσης συζήτησαν προσανατολιστικά για το θέμα και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να έχουμε μια ισχυρή πολιτική συνοχή στο μέλλον. Στις 29 και 30 Μαρτίου του 2011 είχαμε τη συνεδρίαση των διευθυντών των αρμοδίων για την χωροταξική ανάπτυξη και εκεί εγκρίναμε την χωροταξική ατζέντα για το 2020 και στην άτυπη υπουργική συνεδρίαση της 19ης Μαΐου παρουσίασε το ζήτημα η Ουγγρική Προεδρία στους Υπουργούς. Επίσης, 30 Μαρτίου είχαμε στη Βουδαπέστη μια συνάντηση υψηλού επίπεδου για την εδαφική συνοχή και μιλήσαμε για την θεματική συγκέντρωση, την ευελιξία και μια πολιτική συνοχή η οποία θα προσανατολίζεται κυρίως προς τα αποτελέσματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της τελευταίας συνεδρίασης εγκρίθηκε ο διπλός στόχος της θεματικής συγκέντρωσης. Δηλαδή αυτή η πολιτική θα πρέπει να συνδυάζεται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 και τονίζει ότι βασικό στόχο είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Επίσης, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι για να, μία, ε, να έχουμε μία αποτελεσματική ε, πολιτική συνοχή έπρεπε να έχουμε και την απαραίτητη ευελιξία και οι περιφέρειες πρέπει να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυναμικές τους. Τα κράτη-μέλη επίσης υποστήριξαν σαφέστατα ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να στοχεύει στην... στα αποτελέσματα. Χρειάζεται, λοιπόν, πολιτικ... Χρειάζονται πολιτικές για το μέλλον που να βασίζονται στα διδάγματα που είχαμε στο παρελθόν και αυτό όμως χωρίς να αυξηθούν τα διοικητικά κόστη. Επίσης, τους τελευταίους μήνες εργαστήκαμε σκληρά στην ομάδα εργασίας για τις διαρθρωτικές δράσεις στο Συμβούλιο. Και πέρα από το να προετοιμάσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αναφερθήκαμε στα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στο μέλος της πολιτικής συνοχής. Βασικό στοιχείο της Προεδρίας ήταν μια άτυπη συνεδρίαση υπουργών στην Ουγγαρία. Και οι Υπουργοί Χωροταξίας ενέκριναν την ε, PA 2020, την χωροταξική ατζέντα για το 2020. Πρόκειται για ένα στρατηγικό έγγραφο που οποίο καθορίζει ποιο, ποια είναι η θέση της χωροταξικής συνοχής στο πλαίσιο του 2020. Επίσης τονίζει το βασικό ρόλο των μέτρων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ρόλο της πολιτικής συνοχής. Με αυτήν τη νέα ατζέντα εμείς θέτουμε τα θεμέλια της νέας πολιτικής συνοχής, αλλά επίσης ορίζουμε ότι όλες οι πολιτικές της Ένωσης αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Η Ουγγρική Προεδρία για την χωροταξική ατζέντα ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδικασία διαβούλευση σε διακυβερνητικό επίπεδο και στόχος ήταν η επεξεργασία συμπερασμάτων της Προεδρίας. Τα κράτη-μέλη επίσης ε, δέχθηκαν ε, ενιαία ότι οι πολιτικές θα πρέπει να επικεντρώνουν τους στόχους τους και να έχουμε μία ισορροπημένη συνοχή. Επίσης, στις 29 Μαΐου θελήσαμε να πούμε ότι έχουμε μια πολιτική συνοχή η οποία διατηρείται και εμείς δώσαμε προσανατολισμούς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το περιεχόμενο του νομοθετικού πακέτου που θα παρουσιαστεί σύντομα. Θέλω να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο τοποθετήθηκαν λέγοντας ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να συγκεντρώνεται προς τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα και θα πρέπει να δημιουργηθεί κατά συνέπεια να δημιουργηθούν κίνητρα και σε άλλες ε, παράλληλες πολιτικές. Εμείς θεωρούμε ότι η Ουγγρική Προεδρία κατάφερε να ολοκληρώσει τους στόχους της. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προσπαθήσουμε να έχουμε μία κοινή θέση για, για τα στρατηγικά ζητήματα και για να μπορέσουμε να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εμείς αναλύσαμε τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν κατά την εκτελεστική φάση αυτών των πολιτικών. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι εργασίες ετοίμασαν πολύ σωστά την πορεία ούτω ώστε να έχουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε γέρος τα προγράμματα συνοχής μετά το 2013. Και για να ολοκληρώνω θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους αυτή της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλη την υποστήριξη που μας δώσανε κατά την Ουγγρική Προεδρία. Αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έκανε ιδιαίτερα σημαντική τεχνική και πολιτική δουλειά και με την ενεργική τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Προεδρίας συνεισέφερε ιδιαίτερα στις εργασίες μας. Σήμερα έχουμε μια ουσιαστικότητα περίοδο μπροστά μας είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία προπαρασκευής της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Πρέπει λοιπόν εμείς να στροφούμε στη δουλειά. τότε την τελευταία μέρα της Ουγγρικής Προεδρίας κατατέθηκε η πρόταση της Επιτροπής για το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Και σήμερα το πρωί εγώ συνάντησα την κυρία Μπιλκόφσκα και διαπιστώσαμε ότι οι Πολωνοί συναδελφοί έχουν μπροστά τους ένα τεράστιο έργο, διότι πολύ σύντομα η Επιτροπή θα παρουσιάσει το νομοθετικό πακέτο για τις πολιτικές συνοχής βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Συζητούμε αυτά τα νομοθετικά σχέδια μέσω μιας νέας διαδικασίας μέσα στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε ως συμπεράσματα στα, στα συνοπτικά πρακτικά της Προεδρίας να ληφθεί υπόψη. Είναι μια περίοδος με μάτι προκλήσεις. Ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε μια εργασία που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε τους τα κονδύλια με αποτελεσματικό τρόπο και θα υποστηρίξει και τους, ε, την επίτευξη των στόχων ε, της Ευρώπης 2020. Βασιζόμαστε στη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υφυπουργέ Κόβατς. Αυτές τις ευχαριστίες ε, θέλω να τις επιστρέψω. Και εμείς χαρήκαμε ιδιαίτερα με το να συνεργαζόμαστε μαζί σας και γνωρίζουμε τη θέση της θέσης του Συμβουλίου. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο έχουμε και εμείς τις θέσεις μας που καθορίσαμε στις διάφορες εκθέσεις και ενδιαφέρον θα γίνει όταν οι προτάσεις για τον κανονισμό υποβληθούν και όταν θα είναι δεδομένες. Και κατά την τελευταία περίοδο με τους Ούγγρους συναδέλφους στην Περιφερειακή Επιτροπή κάναμε εξαιρετική δουλειά. Τώρα όμως θα δώσω τον λόγο στους συναδέφους. Πρώτος, ο συντονιστής του ΕΛΚ, ο κύριος Φανίστερ Ρόι. Παρακαλώ κύριε Φανίστερ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι ευχαριστώ για το ότι στην μετάβαση από την μία προεδρία προς την άλλη έχουμε αυτή την ευκαιρία να ακούσουμε τις θέσεις της ουγγρικής πλευράς. Έχουν σημειωθεί πρόοδοι και η μεγαλύτερη πρόοδος, πιστεύω εγώ, ότι σημειώνεται στα πιο ενδιαφέροντα χαρτοφυλάκια όταν πρόκειται για τους όρους και προϋποθέσεις που θα υπάρχουν, δηλαδή για την αξιολόγηση όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων και τη χρήση κονδυλίων. Θα πρέπει να αποσυνδεθούν όλα αυτά από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αφενός πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματική η υλοποίηση, η εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά πρέπει να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη. Να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη ώστε πραγματικά να μπορέσουν την οικονομική διακυβέρνηση, την economic governance, να την προχωρήσουν και να πάρει θετική τροπή. Στο Γκέρντελε είχα πάει, αν το προφέρω και σωστά κιόλας, στην Ουγγαρία είχα, ήμουν και εγώ παρόν και με το λεωφορείο πήγαμε στην πρωτεύουσα, την Βουδαπέστη. Και μετά τη συνεδρίαση έπρεπε να επιστρέψουμε αμέσως και παρέμεινα και μια μέρα επιπλέον επιτόπου για να δω τι γίνεται στο ίδιο το Γκέντελε και ο Δήμαρχος ήταν πραγματικά υπερήφανος για το ότι υπήρχαν νέοι δρόμοι, νέοι, ε, νέες οδοί που είχαν δημιουργηθεί και το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη παρουσία εκεί γιατί βρισκόμαστε, οι πιο πολλοί είχαν πάει στην πρωτεύουσα. Είναι λοιπόν σημαντικό σε τέτοιου είδους συναντήσεις ε, να μπορεί κανείς να γνωρίζει και να εξοικειώνεται με την ε, περιφέρεια και την περιοχή. Είχαμε μια μέρα όλοι και όλοι για να δούμε πάσης φύσεως σχέδια και προγράμματα. Με πιο διαφορετικό τρόπο θα έπρεπε να κατανείμουμε τον χρόνο μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πέρα από αυτό πιστεύω ότι η ημερήσια διάταξη, ιδιαίτερα για την περιφερειακή ε, για τα περιφερειακά θέματα και μια νέα συνεργασία. Η περιφερειακή διάσταση προστέθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας ως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει τώρα να ενισχυθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 7% νομίζω. 7% θέλησε να αυξήσει τα κονδύλια και τώρα θα υπάρξει και ένα διαμεσολαβητικό ταμείο, ένα ταμείο διασύνδεσης. 33% συνολικά θα αυξηθούν τα κονδύλια και βλέπω ότι ακολουθούν όλα αυτά χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν από εσάς για να υπάρχει να διασφαλίζεται η ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία. Είναι αποτέλεσμα και της δικής σας δουλειάς και επιρροής αυτό και έχετε πλήρως την υποστήριξή μας γι' αυτό. Μία ερώτηση έχω. Η χρήση των κονδυλίων, η χρήση για στόχους στέγασης, για τη στέγαση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Πριν από δύο ε, χρόνια προσαρμόστηκε, τροποποιήθηκε ο κανονισμός. Και τώρα έχουμε ένα πλαίσιο τρομά τους τσιγκάνους και άλλες στοχομάδες θα μπορούν να γίνουν περισσότερα όσον αφορά τη στέγαση. Παρατηρώ όμω ότι αυτή η προσφορά, αυτή η δράση δεν έχει προαθεί ιδιαίτερα ούτε στην Ουγγαρία ούτε και σε πολλές άλλες χώρες. Στη Ρουμανία για παράδειγμα ή και στην Ουγγαρία πρέπει να πει κανείς ότι αυτή την πορεία, αυτή την κατεύθυνση ξεχωρίζουμε. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Υπάρχει κάποια εξήγηση. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Μέχρι στιγμής η απορροφητικότητα, η διάθεση των κονδυλίων δεν είναι η ιδανική παρότι οι ανάγκες είναι τεράστιες. Σε ευχαριστούμε κύριε Φανίστερ Ρόι και για τους φιλελεύθερους ο κύριος Τόιρα παρακαλώ. Ναι κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα μια εκπροημίου παρατήρηση. Η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε με συζητήσεις και αποσυζητήσεις που συναρτώντουσαν με την ανησυχία μας για την ελευθερία του τύπου στην Ουγγαρία και παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς τη συζήτηση για την συνταγματική αλλαγή. Υπάρχουν αυτά τα μελήματα, αυτές ε, οι ανησυχίες. Θέλω να τα αναφέρω αυτά εκ προημίου και σίγουρα τον ένα ή άλλο συνάδελφο τους έκαναν κάπως να απογοητευθούν όσον αφορά την συνεργασία για παράδειγμα στην περιφερειακή διαρθρωτική πολιτική ή την πολιτική συνοχής σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι την Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου την θεωρούμε πολύ επαγγελματική επαγγελματική με κέντρο βάρους ε, που ακριβώς συζητήθηκε προηγούμενα από μας για τη μακροπεριφερική συνεργασία Εκεί διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο η Ουγγαρία για τη στρατηγική διαπεριφερειακή συνεργασία για το Δούναβι. Σας ευχαριστούμε διότι αυτή η συνεργασία διαπεριφερειακά είναι μια συνεισφορά υπέρ της σταθεροποίησης της Ευρώπης όσον αφορά και τα θέματα μειονοτήτων ε, και αυτά δεν θα διαδραματίζουν ε, κάποιο ρόλο στο μέλλον, θα ξεπεραστούν τα προβλήματα και μέσα σε ένα σφαιρικότερο πλαίσιο που θα αναζωογονηθεί θα διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο ώστε και η Ουγγαρία στο μέλλον σε αυτόν τον τομέα να μπορεί να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό ρόλο. Ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να παρέμβω είναι μια ερώτηση. Αύριο εδώ στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή θα ψηφίσουμε για μια έκθεση για τη δική μου ακριβώς έκθεση που αφορά τα ποσοστά απορρόφησης, απορροφητικότητας των κονδυλίων των διαθροτικών ταμείων. Δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν περιφέρειες που με πολύ καλούς ρυθμούς απορροφούν κονδύλια που τα διαθέσιμα κονδύλια και τους τίτλους ε, τα χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, να προαχθεί η διάχυση γνώσεων και να μπορέσουν οι περιφέρειες να συμμετάσχουν και να καλύψουν τα κενά έναντι άλλων πιο προηγμένων περιφερειών. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν προβλήματα. Θα ήθελα τη δική σας αξιολόγηση. Πώς βλέπετε εσείς ως Ουγγρική Προεδρία το θέμα της απορροφητικότητας κονδυλίων. Ακριβώς επειδή εσείς προέρχεστε από την κυβέρνηση μιας χώρας που την μεταφορά από την μεταβατική περίοδο από την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία της κομμουνιστικής περίοδου προς ένα πιο φιλελεύθερο καθεστώς της οικονομίας της αγοράς αυτή την μετάβαση τη γνωρίζετε καλύτερα. Τι φταίει για αυτή τη χαμηλή απορροφητικότητα, τι θα συνιστούσατε να γίνει για να βελτιωθούν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ συνάδελφε για αυτή την παρέμβαση. Ο συνάδελφο Τάμας Ντόιτς έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, καλό σας απόγευμα. Αν μου επιτρέπετε, και εγώ θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις, σύντομες παρατηρήσεις σε αυτήν την τόσο εξειδικευμένη περιεκτική παρουσίαση που μας δώσατε για τις ε, δραστηριότητες της Ουγγρικής Προεδρίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω κάτι. Να τονίσω ότι στις Ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητούσαμε, συζητήσαμε τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές αυτά τα θέματα και πάντα η συζήτηση αυτή ήταν χαρακτηριζόταν, πώς να το πω, από ένα κριτικό πνεύμα και υπήρχαν και πολλές ε, επικρίσεις και πολλές φορές υπήρχαν και επιθέσεις στην Ολομέλεια κατά της Ουγγρικής Προεδρίας, πιο συγκεκριμένα κατά της ε, Ουγγρικής Κυβέρνησης, από τους πράσινους, από τους σοσιαλιστές και άλλους. Και σε αυτές τις επικρίσεις, πολιτικές επικρίσεις που ήταν και πολλές φορές ε, οξύτερες και που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη με κάποιο ας το πω έτσι πιο επιθετικό τρόπο επειδή η κυβέρνηση αυτή που είχε αναλάβει την Προεδρία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από το έργο το ίδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνει πάντα και το καλό παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα αναφέρθηκε για, σε σχέση με τις δραστηριότητες της καταδεικνύοντας, αποδεικνύοντας ότι σέβεται τις αξίες και τις αρχές της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Αυτό αναφέρθηκε σε πολλές ολομέλειες και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συγχαρώ την Ουγγρική κυβέρνηση διότι παρόλες αυτές τις επικρίσεις και τις επιθέσεις δεν κατάφεραν να παρεκκλίνουν την, Ευρω... Ουγγρική Προεδρία ούτε κατά κεραία από τα όσα είχε παρουσιάσει ο Βίκτορ Όρμπαν κατά την Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Και ακριβώς για την πολιτική πολιτικής συνοχής. Για την πολιτική συνοχής το τελευταίο αυτό εξάμεινο ταυτόχρονα ενώ οδηγούσε σε καλή κατεύθυνση την πολιτική συνοχή ε, η Ουγγρική Προεδρία ήταν σε θέση να αλλάξει πλήρως τις δομές ε, της ε, διαχείρισης της περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να πω ότι η Ουγγρική κυβέρνηση όχι μόνο μπόρεσε να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική και τις πολιτικές συνοχές, αλλά επίσης υιοθέτησε το ότι πρέπει να δίνεται το καλό παράδειγμα παράδειγμα και το έκανε. Έδωσε το καλό παράδειγμα με υποδειγματικό τρόπο όσον αφορά την εσωτερική πολιτική ζωή της Ουγγαρίας. Και αυτό μπορεί να είναι υπόδειγμα για πάρα πολλές χώρες που μπορούν να μιμηθούν αυτό το παράδειγμα. Κατά δεύτερο λόγο στη συνέχεια αναμένω, ελπίζω ότι η επόμενη Προεδρία, η Πολωνική Προεδρία και αυτή θα χαρακτηρίζεται από αυτό το πνεύμα στενής συνεργασίας με το Ευρωκοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα με τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπως κατά τη διάρκεια και της Ουγγρικής Προεδρίας από πλευράς της Ουγγρικής Κυβέρνησης. Αυτού του είδους οι Προεδρίες μπορούν πραγματικά να συνεισφέρουν ώστε να πάψουν και να τερματιστούν οι δια θεσμικές και ιδιοργανικές τριβές και αντιπαραθέσεις που δημιουργούν ανησυχίες στους πολίτες και που δεν μπορούν να κατανοήσουν για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι ιδιοργανικές θεσμικές ε, τριβές και αντιπαραθέσεις. Και το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω όσον αφορά τα όσα μας είπε ο Υφυπουργός για τα αποτελέσματα της Ουγγρικής Προεδρίας σε σχέση με τα διαφορετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και με συνενετικό τρόπο, θέλω να πω ότι συμφωνώ ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες ουσιαστικά συμβαίνει το εξή σαν να, είχαμε, σαν να δημιουργήσαμε ένα αρμονικό χορό βάλς ευρωπαϊκό, έναν ευρωπαϊκό χορό. Ο ρυθμός ε, είναι ικανοποιητικός. Θα ήθελε το Κοινοβούλιο όμως περισσότερα να δαπανώνται για την ε, πολιτική συνοχή. Έρχεται ξαφνικά το Συμβούλιο, λέει όχι, λιγότερα θα πρέπει να είναι αυτά τα κονδύλια. Το είδαμε αυτό με δύο ε, αφορμές φέτος. Έχουμε και τον μελλοντικό προϋπολογισμό του 2012, έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τη δέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι όπως διατυπώθηκε. Το Συμβούλιο όμως θέλει πολύ λιγότερα κονδύλια να δώσει για την πολιτική συνοχή κατά το 2012 από πλευρά προπολογισμού σε σχέση με την αρχική πρόταση του προσχεδίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λαμβάνοντα υπόψη την περίοδο μετά το 2013, να πούμε ότι ακριβώ το Συμβούλιο, το Συμβούλιο ήταν εκείνο το οποίο παρουσίασε συμπεράσματα με προοπτική για την πολιτική συνοχή του 2013 που να συμπίπτουν με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σφιχτόχερο και τσιγκούνικο, είναι εκείνο το οποίο τοποθετήθηκε έτσι. Και τέλος θέλω να διατυπώσω μια ερώτηση κύριε Υφυπουργέ για τους δύο στρατηγικούς στόχους της Ουγγρικής Προεδρίας που είχε προασπίσει το πρόγραμμα πλαίσιο, τη στρατηγική για τους Τσιγκάνους, τους Ρωμά αφενός και δεύτερον την έγκριση της μακροστρατηγικής για την διαπεριφερειακή συνεργασία για το Δούναβι. Πείτε μας κύριε Υφυπουργέ, ποιες προοπτικές υπάρχουν μέχρι το 2020 σε αυτές τις δύο συνιστώσεις. Ευχαριστώ. Okay. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων είναι αυτές βέβαια και επί της ουσίας τελείως διαφορετικοί τομείς καλύπτονται και θίγονται. Και γι' αυτό θα πρότεινα ο κύριος Υφυπουργό καταρχήν να προσπαθήσει να απαντήσει. Παρακαλώ. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, eh, képviselő úrak, akik a kérdés. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου διατυπώσατε. Θα ε, προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αναφύονται σε σχέση με την πολιτική σύνοχη και με την πολιτική, πολιτική περιφερειακή πολιτική για τον συντονισμό για την ανάπτυξη που ανα, ε, ενδιαφέρουν περισσότερο τη δική σας κοινοβουλευτική επιτροπή. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα πρέπει να πω, με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός των ε, βιωμάτων του κυρίου Φαν Νίστερρόι. Αυτή η εμπειρία είναι πολύ σημαντική για μας. Να υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ των πολιτών μας με αυτά τα θέματα. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό εκείνοι που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις να μπορούν να γνωρίζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών επί τόπου, στα χωριά, στις περιοχές, στις περιφέρειες των διαφορετικών κρατών μελών και από πρώτο χέρι να μπορούν να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής και να μπορούν από πρώτο χέρι χέρι να γνωρίζουν τι γίνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο υπό το πρίσμα αυτή τη δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά και υπό το πρίσμα περαιτέρω οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για την εφαρμογή και λειτουργία της πολιτικής συνοχής σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι υπερήφανα για τέτοιο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Κοκομπού θα κάνει επίσημη ε, επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία. Είμαστε απόλυτα στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού για την ανάλυση εκείνων των μιζώνων ε, προγραμμάτων και εγχειρημάτων. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να συλλέξουν από πρώτο χέρι οι ευρωβουλευτές επί τόπου. Επίσης αληθεύει και είναι σωστό όσον αφορά τα θέματα της περιφερειακής ημερήσιας διάταξης, του θεματολογίου της περιφερειακής ανάπτυξης. Όλα τα θέματα που αφορούν την πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική είχαν στενότατη διασύνδεση με την Ουγγρική Προεδρία που όταν θα θυμ, αν θυμόσαστε πέρσι το φθινόπωρο είχαμε μια εικόνα στα μέσα ενημέρωση στα, στον τύπο για την πολιτική συνοχή και μπορείτε να δείτε ότι υπήρξε σημαντική ανάπτυξη ανάπτυξη αυτής της εικόνας. Σημαντική ανάπτυξη που μπορεί να τεκμηριωθεί και με στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν το ότι καταφέραμε να προσαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά το, ε, την αποτελεσματικότητά μας σε σχέση με τη μείωση του ποσοστού σφάλματος έναντι προηγουμένων ετών. Και έτσι αποδείχθηκε ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να συνεισφέρει να επιληθούν πολλά προβλήματα που δημιουργούνται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις περιφέρειές της, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα των συγκάτων Αμερικάνων για παράδειγμα που αναφέρθηκε από διάφορους ευρωβουλευτές. Στη συνέχεια για να απαντήσω συγκεκριμένα πιο χειροπιαστά στην ερώτηση του κυρίου Φανίστερ Ρόι. Είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη που ήδη δόθηκε σε σχέση με την πολιτική συνοχής για την πολιτική ένταξης και ολοκλήρωσης των τσιγκάνων και της ένταξής τους. Είναι πολύ σημαντικό όπως είπε ο κύριος Φανίστερ Ρόι να δεσμεύσουμε και να θέσουμε σε αναλογία τον πληθυσμό πληθυσμό των Ρώμα με τον ευρύτερο πληθυσμό και να δώσουμε και την ε, αντίστοιχη βοήθεια αναλογικά όπως χρειάζεται καταφέραμε να ε, στέψουμε με επιτυχία αυτή την πρωτοβουλία. Για μας αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα, ευρωπαϊκό, ε, ένα ουγγρικό ίδρυμα το οποίο ε, προωθεί την κοινωνική ένταξη και την ολοκλήρωση και αφομοίωση των Ρωμά στην Βουδα, Βουδαπέστη και στην περιοχή του Μπόρσοτ που είναι μία από τις πιο καθυστερημένες περιοχές. Πρόκειται για μια χρηματοοικονομική υποστήριξη startup, εκ ε, άμεση υποστήριξη εκ των κάτω προς τα άνω για να βοηθηθούν οι μικρέ ε, μικρές επιχειρήσεις με μέτρα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης για να μπορέσουν να ενταχθούν κοινωνικά και πολιτικά οι Τσιγκάνοι. Και υπάρχει μια ολόκληρη σειρά διατάξεων που στοχεύουν στο να βελτιώσουν την κατάσταση της ε, μειονότητας των τσιγκάνων. Στη συνέχεια, απαντώντας στο ερώτημα του κυρίου Τόιρα, ο οποίος ανέφερε τη σημασία της δυνατότητας βελτίωσης των ποσοστών απορρόφησης των κονδυλίων, των διαδοτικών και άλλων κονδυλίων από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων από την Ουγγαρία για παράδειγμα. Όμως στο επίπεδο εκτέλεσης σταδιακά μπορούμε να πούμε ότι βελτιωθήκαμε και υπήρξαν βελτιώσεις. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Αν αναλύσουμε όμως τον μέσο όρο σε σχέση με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουγγαρία επιτυγχάνει αυτό το μέσο όρο, τον φτάνει. Και είναι σημαντικό διότι οι δράσεις της κυβέρνησης μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε να γνωστοποιηθούν αυτές οι δράσεις, αυτά τα μέτρα και όλα αυτά συνεισφέρουν ότι ένα από αυτά τα μέτρα ήταν να βελτιωθεί η ταχύτητα και ο ρυθμός και η αποτελεσματικότητα των κονδυλίων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι οι δράσεις έχουν νόημα μόνο όταν μπορούν να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια με ταχύς ρυθμούς για να είμαστε αποτελεσματικοί. Η πείρα δείχνει ότι υπάρχει μια απλούστευση, μια εξαπλούστευση. Και αυτό είναι ένας από τους μαγικούς όρους που είχε χρησιμοποιήσει η Ουγγρική Προεδρία. Simplification, η απλούστευση, εξαπλούστευση η δυνατότητα δηλαδή να βελτιωθούν οι ρυθμοί και τα ποσοστά απορροφητικότητα από τα κράτη-μέλη με απλούστευση γραφειοκρατική και διοικητική. Προσπαθώ τώρα να απαντήσω στον κύριο Ντάιτ. Ο κύριος Ντάιτς αυτά τα οποία ανέφερε είναι δύο μεγάλες επιτυχίες της Ουγγρικής Προεδρίας. Βρισκόντουσαν στο, στο πρόεδρο της Ουγγρικής Προεδρίας και ιδιαίτερα μας ικανοποιεί ότι μπορέσαμε να ε, πετύχουμε τους στόχους στην μακροστρατηγική διαπεριφερειακή για τον Δούναβη και την πολιτική μας υπέρ των συγκάνων. Ξεκινώ για την, με την πολιτική για τη συνοχή. Ήδη προανέφερα κάτι για τον κύριο Φανίστερ Η πολιτική συνοχής πάντα ήταν ευαίσθητη ευαισθητοί, ευαισθητοποιημένοι για τα προβλήματα της μειονότητας των συγκάνων. Προσπαθήσαμε ήδη στο παρελθόν να βοηθήσουμε την κοινωνική του ένταξη, την ένταξη των συγκάνων, της μειονότητας των συγκάνων στην κοινωνία μας. Και έτσι στην περίοδο προγραμματισμού από το 2007 έως το 2013 όταν έρχεται η στιγμή όταν επρόκειτο για την κατάρτιση προγραμμάτων δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή για την ένταξη κοινωνικών ομάδων που είχαν περιθωριοποιηθεί. να ε, θυμόσαστε κυρίες και κύριοι ότι είχε εκπονήσει τέτοιου είδους προτάσεις στο ευρωκοινοβούλιο από κοινού με το συμβούλιο άρα γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. δεύτερον όσον αφορά την στρατηγική πλαίσιο για την ένταξη των τσιγκάνων είναι ένας από τους πυλώνες ε, στην ευρώπη για την ένταξη αυτής της μειονότητας. Είναι τα θεμέλια αυτά και κάθε χώρα θα εκπονήσει δικά της θεμέλια για την ένταξη των συγκάνων. Αυτό που προτείνουμε είναι ένα πλαίσιο λοιπόν. Σε αυτό το πλαίσιο θα διαδραματίσουν ένα μεγάλο ρόλο τα κονδύλια τα οποία θα βοηθήσουν για αυτή την ένταξη. Είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμός στην υλοποίηση των προγραμμάτων και σχεδίων. Πρέπει όμως να υπάρχει και ελαστικότητα όσον αφορά τα κράτη-μέλη, διότι είναι ένα πολύ περίπλοκο σύνθετο το θέμα και πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία σε σχέση με το τοπικό επίπεδο το περιφερειακό επίπεδο, το κρατικό επίπεδο διότι υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές ή συνιστώσεις που αφορώνται ιδιαίτερα όσον αφορά τους Τσιγκάνους. Όχι μόνο έχουμε το θέμα της ένταξης των Ρωμανί, των Τσιγκάνων, πρέπει να βελτιωθεί η ένταξη όλων των μειονεκτικών ομάδων, των μειονεκτούντων ομάδων ή των περιθωριακών ομάδων. Θέλουμε να αποφύγουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να απομονώσει ή να καταστήσει νησίδες την πολιτική για τους τσιγκάνους, για τους φτωχούς, για τους νέους, τους ανήλικους. Γι' αυτό θέλουμε το θεματολόγιο για την στρατηγική του 2020 να συναποτελεί έναν οριζόντιο στόχο για όλες τις εξειδικευμένες πολιτικές. Μετά στη συνέχεια για την υλοποίηση της στρατηγικής ή της μακροστρατηγικής διαπεριφερειακά για τον Δούναβη αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν νέα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτό θα δημιουργούσε δυσκολίες. Μπορώ όμως να σας πω κύριε Ντόιτς ότι στην υλοποίηση από τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη όταν θα η ώρα εφαρμογής αυτών των στρατηγικών θα εξεύρουν τα αναγκαία κονδύλια για να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές. Η συνοχή. Η συνοχή δεν είναι μόνο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να την προσεγγίζουμε ως συνοχή στα τεκτενόμενα στην λεκάνη του Δούναβη. Και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει προφανώς να είναι σεβαστό το επίπεδο της επικουρικότητας και της διαστρωμάτωσης ε, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων. Έτσι να εμπλέκονται οι κυβερνήσεις, αλλά επίσης οι τοπικές αρχές και περιφερειακές αρχές και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτονόητο. Δεν πρόκειται μόνο αποκλειστικά και μόνο για την προσπάθεια να επιλύσουμε προβλήματα, τα οποία είναι βέβαια σημαντικά σε αυτή την μακροπεριφέρεια και διαδοχικά ή σταδιακά όπως είπε ο κύριος Τόιρερ τα σύνορα οι μειονότητες να μπορέσουν να ενταχθούν και να υπερβούμε τα προβλήματα αλλά πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων των κεντρικών κυβερνήσεων, τοπικών κυβερνήσεων, περιφερειακών κυβερνήσεων, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των εμπλεκόμενων ώστε να εκπονήσουμε μια μεθοδολογία κοινή. Αυτό είναι τεράστια σημασία κυρίες και κύριοι και πρέπει να το προσθέσω είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι ότι Ω ως χώρα της λεκάνης του Δούναβη μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συνεργασία με σημαντικό τρόπο. Ευχαριστώ. herzlichen Dank. ευχαριστώ πολύ. Και πάλι εδώ αρχίζουμε τον γύρο ερωτήσεων. Ο συνάδελφος Κέλλη πρώτος, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα και εγώ να, να επενέσω την Ουγγρική Προεδρία για την εξαιρετική της δουλειά για την Ευρώπη και ειδικότερα σε σχέση με τα ζητήματα που μας απασχολούν εμάς, δηλαδή για την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την συνοχή ελπίζω ότι θα μας συνοδεύσει για πολλά από τα επόμενα χρόνια. Σε σχέση τώρα με, το, με την νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης ε, και το Σύνταγμα, κατά τη γνώμη μου διωγγώθηκε αυτό το ζήτημα παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Ε, προφανώς ε, νομίζω ότι ο, Πρωθυπουργός ε, χειρίστηκε πολύ καλά το ζήτημα, εξήγησε ότι έπρεπε να εξηγήσει Είναι γεγονός ότι πολύ συχνά οι πολιτικοί αναγκάζονται να υποκύψουν ε, ε, υπό το βάρος ε, με ανώτερων δυνάμεων. Πρέπει να πω όμως ότι η Ουγγρική Προεδρία τα κατάφερε καλά. Επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές συνεδριάσεις και στο Στρασβούργο και εδώ, θα ήθελα να σας επενέσω για την αφοσίασή σας ε, και κυρίως ε, για ε, τη συνάδελφό σας, την κυρία Γεώργια, δεν ξέρω αν προφέρω καλά το όνομά της, λέει ο μιλητής, γιατί πραγματικά έτυχε ιδιαίτερη κριτικής και παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ συνεπής, ήταν πάρα πολύ ε, συγκροτημένη και είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε επίπεδο ε, προεδρίας, ε, εκπεριτροπής προεδρίας. Η Ουγγαρία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προόδο και, στην, και, για, και για την ίδια τη χώρα αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της εκπεριτροπής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να πω πραγματικά συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ ο κύριος Αγκουράκης έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Ε, καταρχήν μια γενική τοποθέτηση, ένα γενικό σχόλιο. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου ικανοποιημένος και ευχαριστημένος αν στη χώρα μου είχα παρόμοιες συνταγματικές αλλαγές όπως στην Ουγγαρία, αλλά αυτό είναι θέμα του, του γκρικού λαού. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τους Ούγγρους και πρέπει να δούνε πώς θα το αντιμετωπίσουν αλλά δεν πήρα για αυτό το λόγο, για αυτό το, λόγο το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα καταρχήν να σημειώσω ότι από ό,τι γνωρίζω ε, η Ουγγαρία αντιμετωπίζει ακόμα πολύ σημαντικές συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Φαντάζουμε το επίπεδο ανεργίας να είναι αρκετά υψηλό, το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης να είναι αρκετά χαμηλό, ε, άρα η γενική κατάσταση παραμένει δύσκολη αν είχε την καλοσύνη ο κύριος Υπουργό να μας δώσει δύο-τρία στοιχεία που βρισκόμαστε, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας ενδιαφέρει ειδικά ε, που βρίσκεται ο Ουγγρικός λαός. Και μετά από αυτό, δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, ε, αν μου επιτρέψει ο κύριος Υπουργό. Η πρώτη είναι, επειδή και ο ίδιος, επειδή έγινε λόγος και εδώ για το ότι το Συμβούλιο αρνήθηκε την αύξηση τα κονδύλια για, ε, για το πρόγραμμα συνοχής 8,5% πρότεινε το Κοινοβούλιο, 5,5% ήθελε το Συμβούλιο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσε ο κύριος Υφυπουργός να μας πει τα επιχειρήματα του Συμβουλίου στην αύξηση των κονδυλίων για το Ταμείο Συνοχής. Ποια, ποια ήταν τα επιχειρήματα που υπήρχαν, ποιο ήταν το επιχείρημα. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξής αν ε, κατάλαβα καλά, από την τοποθέτηση του κυρίου Υφυπουργού, μίλησε ότι στην εκπόνηση της ε, πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή υπήρχαν αρκετά σημεία συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο προφανώς και ορισμένα ή αρκετά ε, σημεία διαφωνίας των κρατών μελών. Θα μπορούσε να μας πει λίγο πιο αναλυτικά ποια ήταν τα βασικά ζητήματα της διαφωνίας ε, στο θέμα της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις όλες αυτές. Κύριε Μάτουλα, έχετε τον λόγο, παρακαλώ ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τα συγχαρητήριά μου προς την Ουγγρική Προεδρία, όπως το έκαναν και άλλοι συνάδελφοι. Και θα ήθελα να θέσω δύο συγκεκριμένα προβλήματα ε, όσον αφορά τον κύριο Κόβετς. Προέρχομαι από μια περιοχή από την Ανατολική Ρουμανία. Είναι σίγουρο ότι στην Ρουμανία έχουμε προβλήματα απορροφητικότητα κονδυλίων. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην περιοχή από την οποία προέρχομαι εγώ βρισκόμαστε πάνω από το μεσόωρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλεται στις εξαιρετικές σχέσεις συνεργασίας που είχαμε και έχουμε με την Ουγγαρία. Επειδή πρόκειται για την περιοχή Τσόγκρα ε, Μπίχερ έχουμε πολύ καλή διασυνοριακή συνεργασία με την ε, Ουγγαρία και ολοκληρώθηκε ο αυτοκινητόδρομος Όραντ Σέγκεντ και έχουμε και ένα πρόγραμμα για το, την υδροδότηση που θα δώσει δυνατότητα να υδροδοτηθεί και το Μπέκες. Και είχαμε και δύο διασυνοριακά προγράμματα οδών μεταξύ της επαρχίας της Άραντ στην Ρουμανία και της Μπέκες στην Ουγγαρία. Πάνε καλά τα πράγματα όσον αφορά την οδική, τις οδικές υποδομές. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν επικοινωνίες και με, ε, επαφές χωρίς ε, δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας όσον αφορά τον στόχο 3 για την διασυνοριακή συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως όσον αφορά τα θέματα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης όπου στα σύνορα είχαμε τύχη ή είχαμε φραγμούς αξεπέραστους. Ευχαριστώ. Yeah, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτησή σας και τώρα έχουμε κάποια λεπτά, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έτσι λοιπόν τα πάμε καλά από πλευράς χρόνου, αρκετά καλά και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Υφυπουργό για να ολοκληρώσει απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριοι βουλευτές για αυτό το δεύτερο γύρο τοποθετήσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ τους κύριους Κέλλη και Βανίστεροι, διότι φαίνεται ότι τα καταφέρνετε μια χαρά με τα <laughs> με τα ουγγαρέζικα διότι ονόματα όπως ε, Γκένι, Χένι και κλπ δεν προφέρονται και τόσο εύκολα στα ουγγαρέζικα αλλά τέλος πάντων πέρα από το αστείο να σας ευχαριστήσω για, την, για το ενδιαφέρον σας για την εσωτερική πολιτική της Ουγγαρίας και την καθημερινή ζωή στη χώρα μου. Εγώ πιστεύω ότι στα αρμόδια φορά, για παράδειγμα στο, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, σε όλα, σε όλες μας τις δραστηριότητές μας εμείς δώσαμε πάντοτε απαντήσεις και ευχαριστώ και τον κύριο Αγκουράκη για την ερώτησή του και θέλω να σταθώ στην κατάσταση στην Ουγγαρία. Είναι φανερό ότι με και λόγω των προβλημάτων στην Ελλάδα το Συμβούλιο αποφάσισε πολύ σημαντικά ε, πράγματα που αποτελούν ανακούφιση για την Ελλάδα που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει με καλύτερο τρόπο το χρήμα των ταμείων συνοχής και θα μπορέσει η Ελλάδα να ξαναπάρει την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης. Εμείς ε, ακόμη περιμένουμε τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά στην άλλη ερώτηση για τον προπολογισμό του 2012 το Συμβούλιο δεν ενέκρινε την αύξηση Δυστυχώ, αυτή είναι μια απάντηση που σχετίζεται άμεσα και με την οικονομική κρίση που ζούμε αλλά με τα προβλήματα κυρίως που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Όλες οι χώρες προχωρούν σε προσπάθειες εθνικής ε, σταθεροποίησης και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν περιορισμοί για χώρες που θέλουν να μπουν ε, ναι, να έχουν πρόσβαση στα κοινά κονδύλια. Εγώ εύχομαι να τελειώνουμε το νωρίτερο δυνατόν με αυτά τα προβλήματα. Έρχομαι τώρα στην κατάσταση στην Ουγγαρία. Εσείς αναφέρατε ένα σωρό δείχτες και για να σας απαντήσω. Θετικά. Είχαμε θετική ανάπτυξη του συντελεστή ανεργίας και οικονομικοί συντελεστές ε, ε, ισχυροποιούνται κάθε μέρα. Και για να μην σας δίνω μόνο ουγγρικές πηγές, να σας αναφέρω αντικειμενικούς κριτές ή όσα θεωρεί ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί στην Ουγγαρία μεταξύ 3 και 3,5% για το ΑΕΠ είναι πολύ σημαντικό αυτό για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Όλα αυτά χάρη και των καλών εξαγωγών αλλά και των προωθήσεων της κατανάλωσης μέσα στην ίδια την Ουγγαρία. Αυτό το δηλώνει ο Σάιβετα. Έχουμε και την Μπέρντ που λέει ότι θα έχουμε μία αύξηση του ΑΕΠ περίπου 3% και η Ουγγρική κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα μείωσης των δαπανών πολύ σημαντικό. Μπορούμε λοιπόν εμείς να μειώσουμε το έλλειμμα του κράτους από σε 67% και ελπίζουμε να έχουμε σε ένα επίπεδο 70 με 75% το έλλειμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πέρα όμως από τη δημοσιονομική συγκράτηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι καταφέραμε να, να εξοικονομήσουμε πάνω από 10 δις για, την, ε, για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Έχουμε και μεσοπρόθεσμα προγράμματα και μακροπρόθεσμα προγράμματα για τη μείωση του διοικητικού άχθους των επιχειρήσεων. Για τη χρηματοδότηση λοιπόν η Ουγγαρία θα πάει μια χαρά. Επίσης έχουμε και ομολογίες σε δολάρια με διάρκεια 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να λύσουν αυτά τα οικονομικά προβλήματα. Εξού δηλαδή και ο Κινέζος Πρωθυπουργό ήρθε στην Ουγγαρία σε μια περιοδία δηλαδή που έκανε που είχε πάει στο Βερολίνο και στο Λονδίνο και ήρθε στην Ουγγαρία και είπε ότι ήθελε να συμμετέχει στη χρηματοδότηση του χρέους του Ουγγρικού κράτους. Και επίσης η Audi, Opel, η Vodafone και η Ericsson έχουν ε, αρχίσει επενδύσεις πάνω 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουγγαρία. Βλέπετε λοιπόν ότι σε σχέση με τα χάλια των προηγουμένων δύο ετών η κατάσταση πάει πολύ καλά, προχωρούμε πολύ ωραία και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας το λέω εδώ. Και για να απαντήσω και στην ερώτηση του κυρίου Ματούλα, ο, ο οποίος ε, ήρθε στην Ουγγαρία και συμμετείχε στην Ουγγαρία με την Υπουργό Μεταφορών σε μια εκδήλωση όπου εγγενιάσαμε ένα σχέδιο διεθνών συμβάσεων υποδομών για τους ε, κατοίκους των συνόρων με τη Ρουμανία. Έχουμε πολύ ωραίες σχέσεις με τη Ρουμανία. Η Ουγγαρία έχει πολλές όμορες χώρες και επειδή έχουμε και πολλά σύνορα με πολλές χώρες η συνεργασία για μας είναι θεμελιώδης και όπως είπαμε και στο παρελθόν στο μέλλον θα συνεχίζουμε να προωθούμε την εκπλήρωση του στόχου αριθμός 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού σχεδίου έχει κάνει μια πρόταση που τίνει προς αυτήν την κατεύθυνση και θα πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, ε, να ενισχύσει λοιπόν την ε, διασυνοριακή συνεργασία και να βελτιωθεί και η χρήση της δαπάνης. Στο παρελθόν συμμετείχαμε στα EGTC, δηλαδή στις Ευρωπαϊκές Ομάδες Χωροταξικής Συνοχής. Αυτό είναι αρμοδιότητα όμως άλλου Υπουργείου. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω στο όνομα άλλων. Αλλά η Ουγγρική κυβέρνηση προσέχει ιδιαίτερα γιατί θα έρθει η πρόταση της Κομισιόν η οποία θα δημοσιευτεί την 1η Αυγούστου και είναι πολύ σημαντική για τη διασυνοριακή συνεργασία. Ευχαριστώ. Μάλιστα οι ερωτήσεις των συναδέλφων απαντήθηκαν από αυτή την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ, εσάς και την ομάδα σας για άλλη μια φορά για το ότι προσήλθατε εδώ απόψε και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι με τόσο θετικό τρόπο επισκοπούμε τα πράγματα παρότι μπορεί να υπάρχει όπως είναι φυσικό διαφορά απόψεων μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου αλλά τώρα βλέπουμε με θετικό τρόπο, στρεφόμαστε με θετικό τρόπο στα όσα θα ακολουθήσουν και σας ευχαριστούμε θερμά.